Good. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με, την... με τις αλλαγές στη μέση διάταξη. Στο σημείο 8 για την ε, βιωσιμότητα της ε, άγριας πανίδας αυτό θα αναβληθεί. Έχουμε την ε, απόφαση επίσης στις 24 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο να έρθουμε και πάλι σε επαφή με την νομική υπηρεσία. Αυτό θα γίνει αύριο στις 3 αμέσως μετά δηλαδή με τη συνάντηση με τους Εθνικούς Κοινοβουλευτικούς και στη συνέχεια έχουμε τη συζήτηση με τον εισηγητή μας κ. Φάμπριξ για την περαιτέρω διαδικασία στη διαδικασία ΣΥΤΑ. και μετά τα σημεία 19 και 20 σας προτείνω να τα αναβάλουμε, γιατί δεν υπάρχει επαρκής χρόνος. Έχετε κάποιες αντιρρήσεις? Όχι. Ούτως απεφασίστε. Σημείο 2. Πρακτικά. βάσει τη πάγιας πρακτικής. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση η οποία έχει διαβιβαστεί μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας, θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Σημείο 3. Ζωντανά στο διαδίκτυο βγαίνουμε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Οι πολυπληθείς τηλεθεατές μας που μας βλέπουν από τη Λισαβόνα μέχρι τη Λουμπλιάνα, από την Κομοτηνή μέχρι το Βίλνιους και επομένω. Όλα αυτά θα τα δουν οι τηλεθεατές μας. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να είσαστε μετριοπαθείς στον χρόνο αγόρευσης. Επίσης, ήμασταν στο Μπαγκλαντές και έχουμε μια σύντομη έκθεση για τα θέματα αυτά και θέλουμε συμφωνία EGA, Environments Goods Agreements, η οποία βρίσκεται στον 18ο γύρο, θα περατωθεί με μια Υπουργική Σύνοδο 3 και 4 Δεκεμβρίου και δεν θα ήταν κακό να μπορέσουμε εφέτος, εάν γίνει βέβαια κάτι τέτοιο, να έχουμε μια συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου. Σημείο 4. Η κατάσταση των ε, συνεχιζομένων τριγωνικών διαλόγων. Εδώ έχουμε μια πολύ θετική είδηση στις 22 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Υπήρξε επιτυχής κατάληξη της διαπραγμάτευσης για τα λεγόμενα ορυκτά από ζώνες σύγκρουσης, από εμπόλεμες ζώνες. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και τον Ιούλιο, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία για το θέμα αυτό, αλλά και όλη την ομάδα διαπραγματεύσεων. Βλέπω την κυρία Ρένα εδώ. Θέλω να σας συγχαρώ όλους, γιατί νομίζω ότι κατηγάγαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Και έτσι έχουμε καταφέρει να έχουμε δεσμευτική ρύθμιση για μια υπεύθυνη αντιμετώπιση για τέσσερα ορυκτά από το ορυχείο μέχρι το χιτήριο. Και έτσι έχουμε καταφέρει να έχουμε τις καλές, τις σωστές διαδικαστικές ρυθμίσεις. Και είναι καλό λοιπόν να θέσουμε καταρχήν το πλαίσιο για την νομοθεσία με αυτή την απόφαση ώστε να υπάρξει και καλύτερη νομοθεσία για τα θέματα αυτά και αυτό φυσικά ενδιαφέρει πάντα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες. Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας αξιόστροφης πολιτικής εμπορίου. Θα σας δώσω όμως το λόγο αν θέλετε να παρέμετε εδώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρος ότι μου αξίζουν όλα αυτά τα συγχαρητήρια. Θα ήθελα να συγχαρώ όλη την διαπραγματευτική ομάδα, τους και συζητητές γιατί ήταν δύσκολη και πολύ επικοτομητική όμως η συνεργασία μας. Και νομίζω ότι καταφέραμε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία εν τέλει. Μόνο χάρη στην καλή μας συνεργασία, επαναλαμβάνω. Και την ενωμένη θέση της διαπραγματευτικής ομάδας. Ενώπιον του Συμβουλίου. Εν συντομία, Πρόεδρε για τα πρακτικά. Να αναφέρω κάποια από τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας, δεν πρέπει να τα επεξηγήσω ασφαλώς, στην παρούσα φάση να τα αναφέρω καταρχάς σε ό,τι αφορά την υπερχρονική αναφορά των ορεικτών αυτών και κάποιες ε, δεσμεύσεις, πολιτικές δεσμεύσεις, πολύ σημαντικές ε, το οποίο αποτέλεσε και την τελευταία επιτυχία της διαπραγματευτικής μας ε, ομάδας, προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί οι μικρές εξαγωγές δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές αυτές διατάξεις. Ε, έχουμε την αρχή της επιμέλειας, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία όλων των φορέων στην διαδικασία αυτή. Έχουμε τις γραμμές του ΑΣΑ, οι οποίες διέπουν όλη την νομοθεσία και τέλος το Κοινοβούλιο εξασφάλισε σε διάφορες περιστάσεις ότι τα συμπληρωματικά μέτρα θα επιβληθούν προκειμένου να είμαστε ενήμεροι και η Επιτροπή θα υποβάλει τακτικές αναφορές στην, στο Κοινοβούλιο. Το οποίο είναι λογικό δεδομένη τη σημασία ε, τη νομοθεσίας. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τη συνεργασία σα. Ευχαριστώ του συναδέλφου της Επιτροπή. Ε, ευχαριστώ και όλους τους υπαλλήλους για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι ο εισηγητής παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία αυτή, γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερως. Μετά λοιπόν τη συμφωνία της 22ης Νοεμβρίου, το Συμβούλιο στις 7 Δεκεμβρίου θα συζητήσει τα θέματα αυτά στα πλαίσια του Κορεπέρ και ελπίζω ότι το Συμβούλιο να αποτεχθεί το αποτέλεσμα αυτό. Η Προεδρία του Συμβουλίου ουσιαστικά έχει την εξουσία για να ψηφίσει τη συμφωνία. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Έχουμε δει πρόσφατα το παράδειγμα των στατιστικών στοιχείων εξαγωγών, όπου πετύχαμε συμφωνία στο τριμερή διάλογο, αλλά δεν επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα αυτά το Συμβούλιο. Ε, το απευχόμεθα αυτό. Και ελπίζουμε ότι το Δεκέμβριο θα υπερψηφιστεί στο Συμβούλιο το αποτέλεσμα των τριμερών διαλόγων. Θα αποσταλεί στη συνέχεια επιστολή, επιβεβαίωση της συμφωνίας προκειμένου να συνεχίσουμε και εμείς τις διαπραγματεύσεις μας. Ίσως ε, να το ψηφίσουμε το Γενάρη στην Επιτροπή μας και μετά ε, στην Ολομέλεια και στο πρώτο τρίμηνο του 2017 να ολοκληρωθεί αυτή η νομοθεσία. Ελπίζω λοιπόν, να επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμβολή της νομοθεσίας αυτής και ότι αυτά αποτελούν ε, α, μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά τις, ε, τα θέματα διεθνούς εμπορίου. Μάλιστα. Ας περάσουμε στο σημείο 5 τώρα. Αντιπροσωπεία ad hoc στο Παγκλατές. αποφασίσαμε συνάδελφοι να στείλουμε στο Βαγκλαντές μια διαρευνητική αποστολή. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κλωστοϊφαντουργικά. Το Μπαγκλαντές ε, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγό σε παγκόσμιο επίπεδο για τα κλωστοϊφαντουργικά. 85% οι εξαγωγές του Μπαγκλαντές ε, στηρίζονται στα κλωστοφυπουργικά. Και μεγάλο ποσοστό αυτό πάει στην Ευρώπη. 65%. Είναι λοιπόν ο βασικό ε, εμπορικό εταίρο σε θέματα κλωστοϊφαντουργία του Μπαγκλαντέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένη δε τη ε, σημασία, τη οικονομική σημασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και των προβλημάτων από την άλλη που εμφανίζονται διαρκώ ό,τι αφορά την ασφάλεια τη εργασία, προστασία από πυρκαγιέ, δικαιώματα Διαπιστώσαμε λοιπόν στη διάρκεια τη αντιπροσωπεία ε, διάφορα στοιχεία. Καταρχάς, ό,τι αφορά θέματα εφαρμογή του Global Compact για την αντιμετώπιση τη ε, τραγωδία Άνζα Πλάζα. Είδαμε τι βήματα ε, έγιναν προκειμένου και στο μέλλον να είναι διαφορετικές οι συνθήκες που επικρατούν στο Μπαγκλαντές. Είναι λοιπόν σημαντική η χρονική στιγμή. Αυτό αφορά ασφαλώ τι ευρωπαϊκέ εταιρείε και τι ε, λοιπέ εταιρείε ε, που έχουν εμπορικέ σχέσει με την περιοχή του Μπαγκλατέ. Σκοπός μα είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθήκων και ω εκ τούτου λοιπόν συζητήθηκε το θέμα της συμφωνίας με τον Υπουργό Εργασία και τον Υπουργό Εμπορίου. Επισκεφθήκαμε και δύο εργοστάσια. Ένα το οποίο είχε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ό,τι αφορά τα εργασέκα και άλλο ένα εργοστάσιο το οποίο Ε, πέρασε από επιθεώρηση και προτάθηκαν μέτρα βελτίωση. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδο του γεγονό ότι πέρασαν από επιθεώρηση 1.700 εργοστάσια και τελικά καταλήξαμε σε, μια, σε ένα σχέδιο. για την βελτίωση των όρων των ε, ηλεκτρικών ε, εγκαταστάσεων, της ε, στατικής, της δομικής, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 1.700 εργοστάσια είναι μια καλή αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αρκεί αυτό. Όταν θα εκπνεύσει αυτή η συμφωνία, γιατί θα εκπνεύσει το 2018 μετά από πέντε χρόνια, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια διαφορετική συμφωνία με τον Μαγκλαντέ, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίε προ την κατεύθυνση αυτή. Φυσικά. Συζητήσαμε και με την ε, κυβέρνηση των Παγκλαντέ και με την κοινωνία των πολιτών σε ό,τι αφορά τη συνολική κατάσταση, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και πρέπει να σα πω ότι πιστεύω ότι κυρίω τα συνδικάτα είναι ο καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Και γι' αυτό λοιπόν η αλλαγή τη σχετική νομοθεσία για τα εργασιακά στο Μπαγκλαντέ ήταν καθοριστική, προκειμένου να ιδρύεται με μεγαλύτερη ευκολία τέτοια συνδικάτα. 7.200 είναι αυτή τη στιγμή τα συνδικάτα στον Παγκλαντές. Επαναλαμβάνω, 7.200 τα οποία σε κάποιε περιπτώσει οργανώνονται ανά εταιρεία. Και μόνο στην κλωστοϊφαντουργία έχουμε 30 ενώσει τέτοιων συνδικάτων. Παρ' όλα αυτά, παρά τι αλλαγέ αυτέ, ε, μάλλον η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπω. Αυτό που ήταν επίση σημαντικό κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μα ήταν το εξή ότι από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση στο Παγκλαντέ θέλει να δημιουργήσει όσο πιο πολλέ ζώνε εξαγωγή γίνεται 9 έως τώρα. Υπάρχουν θέλουν ε, να, ιδρύσουν 100 για να προσελκύσουν ε, αφενός τους αλλοδαπούς επενδυτές και αφετέρου να βελτιώσουν την παραγωγή τους για προσεξαγωγή. Με μία μικρή υποσημείωση ότι εδώ δεν ισχύει η εργασιακή νομοθεσία. Και αυτό ασφαλώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ταχτούμε. Κλείνοντας, συζητήσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, το τι θα συμβεί αν το Παγκλατές προχωρήσει προς την οικονομική ανάπτυξη και αναπτυχθεί τόσο που τελικά δεν θα θεωρείται λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα. Less developed state. Ξέρετε ότι ε, στις περιπτώσεις αυτές ισχύει ελεύθερη πρόσβαση σε αγορές χωρίς ε, δασμούς, εκτός από τα όπλα, ε, και σε αυτούς τους τομείς ε, συγκαταλέγεται και η κλωστή φαντουργία. Τι θα γίνει λοιπόν, αν βελτιωθεί τόσο η οικονομική κατάσταση του Παγκλαντές που δεν θεωρείται πλέον λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα μπει στο GSP Plus και θα πρέπει να επικυρωθούν 27 τέτοιες συμφωνίες και θα πρέπει την περίπτωση αυτή να γίνει αυτό, το, όχι το 2021, αλλά τώρα ήδη. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα τα εργασιακά. Δεν είναι απλό βέβαια. Γιατί πέρα από το θέμα της ε, βελτίωση τη εργασιακή ε, νομοθεσία και των εργασιακών δικαιωμάτων, μιλάμε και για ανθρώπινα δικαιώματα. Ελευθερία έκφραση. Η ελευθερία έκφραση λοιπόν στον Παγκλαντέ ε, είναι ένα θέμα που μα απασχολεί. Μεγάλα προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει κυριαρχία στην παρούσα φάση ενό κόμματο. Οι διάφορε απόψει καταπιέζονται και ανάλογοι είναι οι περιορισμοί που επιβάλλονται. Άρα και εδώ θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Προκειμένου να καταλήξουμε σε μια σωστή κατάσταση, σε περίπτωση που χάσει το καθεστώς της λιγότερης, λιγότερο αναπτυγμένης χώρας και θέλει να περάσει το JSP. Άλλοι να βλέπουν θετικά τα πράγματα, αλλά αρνητικά βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν είναι εντελώ γεμάτο το ποτήρι. Και όπω ε, λέμε πάντα, εμεί αυτό που θέλουμε είναι προ το συμφέρον ε, του λαού του Μπαγκλατέ να είναι γεμάτο το ποτήρι και να χρησιμοποιήσουμε τη μόχλευση των ε, εμπορικών ζωντημάτων για να βελτιωθεί η εργασιακή νομοθεσία και η λοιπή νομοθεσία. Ήταν, θεωρώ, πολύ εντατική και ενημερωτική η αποστολή αυτή. Θα ήθελα ιδιαίτερως να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Αποστολή στο Μπαγκλαντές, η οποία συνόδευσε πάρα πολύ ενεργά την αντιπροσωπεία μας, μας υποστήριξε πάρα πολύ καλά και μεταξύ άλλων φρόντισε και για την ασφάλειά μας, προκειμένου να φτάσουμε πάλι στο και βλαβής. Εδώ. Αυτά, εν συντομία. Η αναφορά της επίσκεψης σχετικά μάλλον η αναφορά της επισκέψης στον Παγκλαντές. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις να κάνετε. Ίσως και αυτοί που συμμετείχαν στην αποστολή. Δεν θέλετε να είναι έτσι. Δεν θέλει κανένα να λάβει το λόγο. Μπορούμε να περάσουμε το σημείο αυτό και θα υπάρξει όπως ε, ήθιστε μία γραπτή αναφορά σε σχέση με την αντιπροσωπή αυτή. Πάμε στο σημείο 6 τώρα. Hm. Έχουμε προτρέξει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είχαμε πει χθε στι 3.30 ότι θα συζητήσουμε αυτό το σημείο. Κάνουμε ένα διάλειμμα, θέλετε, 5 λεπτών. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt gehen wir weiter in unserer Arbeit. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την εργασία μας. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως με το σημείο 6, να γυρίσουμε στο σημείο 1. Είχαμε αποφασίσει ότι αύριο στις 3 η ώρα θα είχαμε την συνάντηση με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Αλλά μου είπανε μόλι ότι αύριο στις 3 η ώρα δεν θα έχει τελειώσει, δεν θα έχει περατώσει τη γνωμοδότησή της η νομική υπηρεσία, τότε δεν έχει και πολύ νόημα να συζητήσουμε με την νομική υπηρεσία. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι να αναβάλουμε και αυτό το σημείο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, που είναι η επόμενη συνεδρίασή μας, ώστε η αυριανή η ημερήσια διάσκεψη. Θα ξεκινήσει με την ε, ανταλλαγή απόψεων με τον συντονιστή μα και τα υπόλοιπα σημεία στην ημερήσια διάταξη που είπα προηγουμένως 19 και 20 μπορούν να παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη. Έχετε τώρα κάποια αντίρρηση για αυτή την εκ νέου αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Μπίχνερ έχει το λόγο. μήπως θα ήταν δυνατό να έχουμε τουλάχιστον το προσχέδιο της έκθεσης της νομικής υπηρεσίας, οπότε τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Ναι, ναι, αυτή ήταν και η άποψη πολλών άλλων. Αν μπορέσει λοιπόν η νομική υπηρεσία να το κάνει αυτό, αν υπάρχει κάποιο κείμενο το οποίο είναι γραπτό και μπορεί να μας το δώσει, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε ξαλάξαμε και πάλι τη μέση διάταξη και την ξαναεγκρίναμε και αύριο τότε θα έχουμε αυτήν την ε, ανταλλαγή απόψεων, όπως είπαμε, τον συγητή μας και τα υπόλοιπα μια της μέσης διάταξης. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 6. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάπως ιδιότυπο, αλλά και ξεχωριστό σημείο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που το συζητούμε έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με νέους Ευρωπαίους και νέες Ευρωπαίες και να ακούσουμε τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη το Μάιο στο Στρασβούργο είχαμε τη μεγάλη αυτή ε, συνδιάσκεψη με την, ε, που οργανώθηκε από το European News με παρουσία 5.000 νέων οι οποίοι συζήτησαν για τα θέματα της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής και φυσικά αυτό περιλαμβάνει και την πολιτική εμπορίου της ευρωπαϊκής ε, πολιτική εμπορίου του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μας. Και τα απορίσματα αυτής της συζήτησης θα τα μοιραστούν τώρα μαζί μας, με την Επιτροπή μας. Στις 6 ε, Σεπτεμβρίου πήραν όλοι οι συνάδελφοι ένα κείμενο, όπου αναφέρονται τα απορίσματα αυτά της συζήτηση που έλαβε χώρα 50 ιδέες για μια καλύτερη Ευρώπη, ένα καλύτερο μέλλον στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και επομένω υπήρξε και κατά κάποιο τρόπο η προετοιμασία για τη σημερινή συζήτηση. Αυτή η συζήτηση γίνεται και σε άλλες επιτροπές βέβαια, όχι μονάχα σε εμάς αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τους νέους σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχουμε τρεις εκπροσώπους μαζί μας, αλλά δεν είναι αυτό μονάχα. Έχουμε ένα πίνακα τιτιβίσματος με τη χρήση του Twitter και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε διάδραση και να βλέπουμε και σχόλια από τον έξω κόσμο τα οποία θα βλέπετε στον πίνακα. Και η μικρή αυτή η μήνυ ο, ο ακρόασή μας έχει να κάνει με το θέμα δίκαιο εμπόριο, fair trade και επίσης τα θέματα της ε, TTIP. Είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για μας και την Επιτροπή μας. Και έχουμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο που θα μπορέσουν οι νέοι να μας παρουσιάσουν ιδέες οι νέοι αυτοί και εμείς μπορούμε να τα σχολιάσουμε, να ξεκινήσει έτσι μια συζήτηση και γι' αυτό η ιδέα, μάλλον ο στόχος είναι να ακούσουμε από κάθε νέο δύο προτάσεις και αυτές οι δύο προτάσεις μετά θα τύχουν συζήτησης και σχολίασης από εμά, θα τις εγκρίνουμε, θα τις απορρίψουμε, εν πάση δεν έχει σημασία. Έχουμε αρκετό χρόνο τώρα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και έχουμε επίση και την ευκαιρία να υπάρξουν αυτόρμητες παρεμβάσεις, αλλά μόνο τούτο Πιστεύω ότι ο καθένας στο χρόνο αγόρευσής του θα έπρεπε να προσπαθήσει να συγκεντρώσει αυτά που θέλει να πει σε δύο λεπτά μονάχα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα όσο το δυνατόν περισσότεροι να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Οπότε στρέφομαι προς τους ε, τρεις νέους μας, θέλω να τους παρα, παρουσιάσω. Είναι η κυρία Βέντιλ Βίλιαμς, που είναι εδώ, δεξιά. Καλώς ήλθατε. έχει διπλή υπηκότητα, Ηνωμένο Βασίλειο και Τρίνιντατ και Πάκο και είναι ειδική στην, ε, στις πολιτικές επιστήμες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα θέματα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ και επίσης έχει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα από το King's College στο Λονδίνο και έχει αποφυτίσει επίσης και από το Κολέγιο της Ευρώπης στην Βρύγη. Αυτά λένε τα σημειώσει μου. Αυτό λέει. Και καλώς ήρθατε λοιπόν και θερμά, θερμά σας υποδεχόμαστε. Δίπλα είναι ένας ε, φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στη Βιέννη και από την σχολική ηλικία έχει ασχοληθεί με τα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής και υπήρξε και πρεσβευτής εκπαίδευσης των νέων και έχει και εμπειρία στα θέματα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ιδίως στην Αυστρία αλλά και αλλού. καλώ ήρθατε λοιπόν. Αυτή είναι η κυρία Ραμπ, η Δεσπής Ραμπ και μετά έχουμε τον κύριο Τόχ, Τόχβερ, ο οποίος είναι πέντε πέμπτου έτου φοιτητής ιατρικής και ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για τα θέματα υγειονομικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδίω για το πώς μπορούμε να συνδέσουμε την φύση και το εμπόριο, αλλά και την υγεία. Και έχει εξετάσει τα θέματα αυτά με την ε, οπτική γωνία της φύσης, της υγείας, αλλά και της TTIP. Και επίσης είπε ότι είναι ενεργός στην ε, ε, Εστονία για, την, ε, για τον αγώνα της κοινότητας ΛΟΑΔ. και είναι περιφερειακός διευθυντής της Ένωσης Φοιτητών Ιατρικής. Καλώς ήλθατε λοιπόν κύριε Τόχφερ. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο, τις πρώτες ιδέες έχουν να κάνουν με το θέμα του δικαίου εμπορίου. Αυτό θα είναι το πρώτο κομμάτι της ακροασής μας. Και καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ελένα Ραμπ για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας προτείνω ε, να επιβάλλεται έναν υποχρεωτικό δεσμευτικό νόμο για τις ε, ε, βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει αυτές δε οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι υπεύθυνε για όλη την διατροφική αλυσίδα και τα στάθειά της. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει δεσμευτική νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι εθελούσιο σύστημα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE ε, πιστεύουμε επίσης ε, ότι ήρθε η ώρα να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί η ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμης ε, έχει αυξηθεί και είναι πάρα πολύ μεγάλη τα τελευταία, παιδιά, τα τελευταία χρόνια, του δε μεταξύ των νέων παιδιών. Επίσης, η παραγωγή ορισμένων προϊόντων, όπως ας πούμε του κακάο ή του καφέ, έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εργαστεί μαζί τους έτσι ώστε το δίκαιο εμπόριο, το fair trade, ε, να ε, λάβει χώρα και στις περιπτώσεις ε, όλες αυτές και έτσι ώστε να επιτύχουν οι παραγωγοί υψηλότερες τιμές. Είναι αλήθεια ότι δεν ε, ε, είναι όλοι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω έτσι ώστε να έχουν αυτή την επιλογή του, ελευθέρου του δικαίου εμπορίου. Ωστόσο, περισσότερα θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά ε, και να έχουν καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής αλλά και να έχουν και μια καλύτερη ανταπόκριση όσον αφορά την προσέγγιση τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να, ε, ε, να καταλάβουμε ότι το σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα, δηλαδή της εθελούσιας αγοράς ενδεχομένως προϊόντων που να προέρχονται από το ε, δικαίο εμπόριο, δεν είναι μακροπρόθεσμα ε, καλή επιλογή γιατί δεν παράγει μόνιμα αποτελέσματα. Οι μόδες αλλάζουν, οι συνήθειες αλλάζουν και επομένως δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε μόνο σε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της διατροφική αλήθεια. ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ σαφέ το μήνυμά σας. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόμα. Εγώ έρχομαι ενώπιόν σας με μια νέα αντιμετώπιση της ε, ε, παγκοσμιοποίησης. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν μοναδικά πρότυπα και όχι διπλά και να ισχύουν για όλους. Αυτό που σας ζητώ είναι ε, ε, τρία πράγματα. Ε, θέλω και ζητώ από εσά να υπάρχει μία, ένας κώδικας δεοντολογίας ο οποίος θα συνοδεύεται και από συγκεκριμένα πρότυπα και που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής και προμήθειας. Δεύτερον, ε, ε, οπουδήποτε και αν και εφόσον υπάρχει ήδη τέτοιος κώδικας, να διασφαλιστεί η, η παρακολούθηση, ο σεβασμό μάλλον αυτού του ε, κώδικα δεοντολογίας, γιατί βλέπουμε ότι τα σημάδια είναι ιδιαίτερω ανησυχητικά. Τρίτον, πιστεύω ότι θα πρέπει να κατεβληθούν προσπάθειες έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μην εξωθηθούν εκτός εκτός ε, της ε, αγοράς ε, εάν και εφόσον επιλέξουν την πιο δύσκολη οδό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη και να αναφερθούν τέτοια στοιχεία στις εμπορικές συμφωνίες. Όσον αφορά τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγώ θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι συμπεριλαμβάνονται αυτές οι αρχές σε όλες τις συμφωνίες, γιατί από όσο γνωρίζουμε, ακόμα και όταν υπάρχουν ε, τέτοιε υποχρεώσει στι εμπορικέ συμφωνίε, αυτέ ε, δεν ε, εφαρμόζονται. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ακόμα και να εκδιωθούν χώρε εάν δεν εφαρμόζουν του σωστού κανόνε δικαίου εμπορίου. Πολύ ωραία μα, τα είπατε κι εσεί, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ σαφές το μήνυμα και το δικό σα. να δούμε εάν οι συνάδελφοί μου θέλουν να αντιδράσουν. Um, Μιλώ πρώτο εξ ονόματο του ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ιδέε που μα παρουσιάσατε. Σε δύο λεπτά δεν μπορώ να απαντήσω σε όλε τι ιδέε ε, που ακούσαμε. Αυτό που θεωρώ ότι είναι γενικώ ε, σημαντικό είναι αυτά που είπε ο κύριος Ατόμπε για την παγκοσμιοποίηση. Να σας διαβεβαιώσω ότι η διαμόρφωση τη παγκοσμιοποίηση, αγαπητοί νεαροί συνάδελφοι, είναι κάτι το οποίο μα απασχολεί ιδιαίτερα εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η διαμόρφωση τη παγκοσμιοποίηση τι σημαίνει ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε και το ευρωπαϊκό αυτό, την ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία, το, την εκδήλωση I. Μιλάτε για το βιώσιμο μέλλον, για τις θέσεις απασχόληση, Χρειαζόμαστε λοιπόν υπεύθυνη οικονομία, αλλά χρειαζόμαστε και η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ε, μιλάμε για διαμόρφωση της παγκοσμιοποίηση, καταλαβαίνετε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά κανόνες, νομοθεσία, αλλά αφορά και την ήπια εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. την προώθηση σε όλο τον κόσμο των αξιών μας, τον αγώνα για τις αξίες μας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα για να προωθήσουμε τις αξίες μας. Χρειαζόμαστε εταιρική σχέση με την ε, οικονομία. Δεν μου αρέσει να ακούω ιδέες εξαναγκασμού των επιχειρήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξαναγκάσουμε τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα, να δώσουμε εκπαίδευση, κατάρτιση, να δώσουμε κίνητρα. Να πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και επιχειρήματα. Πώς θα φαίνονταν τα νέα αν οι επιχειρήσει έλεγαν θα πρέπει να εξαναγκάσουμε τους νέους ανθρώπους να μάθουν κάτι. Καταλαβαίνετε, ο εξαναγκασμός δεν είναι καλή ιδέα. Αλλά η προάσπιση των αξιών μα είναι καλή ιδέα η διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι ανισότητες, οι βαθιές ανισότητες να αμβληθούν. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τις εξαλείψουμε εντελώς, να τις αμβλύνουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αρένα. Ευχαριστώ πρόεδρο. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Βάλτε τα ακουστικά σας. Vous pouvez Μπορείτε να καταλάβετε ότι μεταξύ μας έχουμε διαφορετικές διστάμενες απόψεις και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που είπε ο συνάδελφος Βίγκλερ ότι δεν έχουμε δυνατότητα να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις να σεβαστούν κάποιους κανόνες. Εξάλλου, την προηγούμενη εβδομάδα καταφέραμε να περάσουμε ακριβώς ε, νομοθεσία ε, η οποία αφορά την ιχνηλασιμότητα των ε, μεταλλευμάτων και που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να κάνουν κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Βίγκλερ που γνωρίζει καλά την έκθεση ως συγητής, πετύχαμε με μεγάλη προσήλωση και προσπάθεια. Και πλέον ε, έγινε υποχρεωτικό ε, το πλαίσιο το οποίο ήταν ε, παλιότερα σε εθελούσια βάση, αυτό που ο ΣΑ ονόμαζε δέουσα επιμέλεια, due diligence. Ναι, κοιτάξτε, είναι σαν να σου λένε καλό θα ήταν να τρέχεις με 130 130 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο ε, υπάρχουν οδηγοί που σέβονται το όριο, άλλοι που δεν σέβονται. Επομένως, το ίδιο με τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες σέβονται και άλλες οι οποίες δεν σέβονται και μάλιστα δεν πρόκειται ποτέ να σεβαστούν οποιαδήποτε ε, αρχή και οποιοδήποτε κανόνα και συνήθως αυτές είναι και οι χειρότερες. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχουν δεσμευτικές υποχρεώσεις. Ε, χαίρομαι που σας ακούω. Είστε μία ε, γενιά η οποία ζητά αξίες, τις απαιτεί και υπεραμείνεται των αξιών αυτών. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει το αίτημα αυτό το οποίο έρχεται και από αλλού, όχι μόνο από τους νέους και πιστεύω ότι ε, όταν λέμε ναι για ε, καλύτερη οικονομία, ανάπτυξη κτλ. Αλλά όταν λέτε shaping the globalization, δηλαδή όταν ε, λέτε ότι πρέπει να προσέξουμε τι μορφή θα δώσουμε στην παγκοσμιοποίηση, αυτό πραγματικά με ικανοποιεί. Χαίρομαι πάρα πολύ και με αγαλίαση ακούω τις παρεμβάσεις σας. Όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, θα, ξέρετε ότι θα συζητήσουμε το θέμα με τον Καναδά, αλλά συζητήσαμε και ε, εμπορικέ σχέσεις με την Αφρική. Ε, υπάρχει ένα κεφάλαιο ε, στις ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών που δεν καταφέρνουμε να περάσουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε και ε, ε, ας πούμε από την πλευρά των Αφρικανών εταίρων. Αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να το περάσουμε γιατί δεν βάζουμε αρκετή πολιτική βούληση. Εάν εσείς λοιπόν είτε μας πρόχνετε, είτε μας κλωτσάτε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, καλό θα μας κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω, λέει ο κ. Μπίχνερ, την ιδέα να έχουμε μια μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων με νομοθετικά μέτρα, ιδίω ό,τι αφορά την τήρηση του δικαίου εμπορίου. Αλλά γνωρίζουμε παράλληλα ότι ιδίω στην Αφρική η παραγωγή του καφέ, του κακάο κτλ. πολλές φορές έχουν ένα ή δύο συνομιλητές εμπορικούς διαπραγματεύονται μονάχα με ένα, μία ή δύο εταιρείε, οι οποίε ουσιαστικά μπορούν να καθορίσουν τι τιμέ που παίρνουν οι καλλιεργητέ. Μήπω λοιπόν, είναι να έχουμε κάποιε συνεταιριστικέ οργανώσει των ε, παραγωγών ή να έχουμε κάποιε τιμέ που καθορίζονται από το κράτο. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό και για τα τρόφιμα. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κατεπηγόντω κάποια ρύθμιση στα θέματα αυτά. Ε, ευχαριστώ και εγώ γερμανικά θα μιλήσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι μαζί μας, γιατί με την επαφή αυτή μπορούμε να ακούσουμε τις απόψεις τους, τις κριτικές τους, τις επιθυμίες τους. Και εγώ χαίρομαι που βλέπω τους νέους οι οποίοι είναι τόσο ενεργοί για τα θέματα του δικαίου εμπορίου. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο εδώ οι άνθρωποι ως καταναλωτές όταν αγοράζουν κάτι να σκέφτονται και από πού προέρχεται. Μήπως υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο είναι υπερβολικά φτηνό, όπως είπε και η Μαρία. Αυτό είναι ένα θέμα, όπως και στην περίπτωση των ε, ορυκτών που προέρχονται από εμπόλεμες ε, ζώνες, να έχουμε κάποια ρύθμιση, να ξεπεράσουμε την εθελοντική μονάχα ρύθμιση. Θα ήταν πολύ ωραία να γίνονται όλα εθελοντικά, αλλά πρέπει εμείς να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο να είναι πιο δεσμευτικό. Και τώρα πρέπει να μιλήσω και για το κοινωνικό dumping. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν υπάρχει ένα ενίο ορισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση του τι αποτελεί το κοινωνικό dumping, αλλά έχουμε όλοι στο μυαλό μας περί τίνος πρόκειται και επομένως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά πόσο οι άνθρωποι παίρνουν μια δίκαια αμοιβή για την εργασία τους και για τις υπηρεσίες που ε, παρέχουν, δηλαδή να έχουμε πέρα του δικαίου εμπορίου στο μυαλό μας και την ανάγκη αξιοπρεπούς και καλά αμοιβόμενης εργασίας. Επίσης, ένα τρίτο στοιχείο είναι το στοιχείο της καταναγκαστικής εργασίας και φυσικά της εργασίας των παιδιών, της παιδικής εργασίας. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και αυτά είναι εξίσου σημαντικά με τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει να είναι στοιχεία τα οποία εμείς τα έχουμε πάντα στις συμφωνίες μας και είναι ακριβώς αυτά τα οποία μας υποδεικνύουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και είναι αυτά τα οποία επιθυμούν και οι πολίτες μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξουν και κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι θα είναι ελεγκτικοί χαρακτήρες. Δεν φτάνει να γράφονται όλα αυτά στις συμφωνίες, πρέπει να υπάρξει και ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας. Δεν έχει νόημα λοιπόν να αποφασίσουμε και να γράφουμε πράγματα τα οποία στη συνέχεια δεν εφαρμόζονται. Αυτό κάνει απαραίτητες και τις κυρώσεις ώστε να υπάρξει και κάποια στεναρότητα στην τήρηση των κανόνων. Είναι πάρα πολλά λοιπόν όλα αυτά τα οποία έχει να κάνει κανείς και γι' αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμες οι ιδέες, Χαίρομαι για όλα αυτά που μας είπατε και σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε αυτά τα οποία κάνετε ήδη. Κύριε Σόλτ, και εγώ να ευχαριστήσω και εγώ θα μιλήσω γερμανικά και εγώ να καλωσορίσω το γεγονό ότι ήρθατε στην Επιτροπή μα. Πολλά είπαν ήδη συνάδελφοι και εγώ είμαι υπέρ των ε, συνθήκων πλαίσιο. Δηλαδή στι εμπορικέ συμφωνίε δεν μιλάμε μόνο για ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Το θέμα είναι και το πώ παράγονται και ε, εξαγάγονται και συνδέονται με τι βιωτικέ συνθήκε του κόσμου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Εκεί είναι ο γρίφος. Τα πρότυπα, οι προδιαγραφές, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο καταφέραμε να το πετύχουμε μετά από αγώνες. Τι γίνεται όμως με τις ικανότητες, τις δυνατότητες μάλλον και τις συνθήκες που επικρατούν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Σε ό,τι αφορά το TTIP, το ΣΕΤΑ ισχύει αυτό. Αλλά Αυτά έχουν σημασία και για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ήπειρο. Πού διαπραγματεύεται συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Είναι συγκεκριμένα λοιπόν ερωτήματα και ζητήματα αυτά. Κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη α, ανταλλαγή όρων ή μήπως θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες αυτές και παράλληλα να αναπτυχθεί η μηπως θα πρεπει να δωσουμε ευκαιρια βιωσιμης αναπτυξη στις χώρες αυτές προκειμένου να μην υπάρχει μόνο ανταλλαγή πρώτων υλών. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος μελητής. Κοιτάξτε. Ε, όταν ήμουν γονέας δεν τα συζητούσαμε αυτά τα πράγματα. Έτσι όπως είχε όμως τώρα η κατάσταση, καταλαβαίνω ότι επικεντρωνόμαστε σε δεντολογικές αρχές. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν διακρίσεις μεταξύ των προδιαγραφών, όπως για παράδειγμα οι προβλητικές προδιαγραφές. Εδώ μπορούμε να καταρτήσουμε νομοθεσία, αλλά όταν πρόκειται για θέματα ανακατανομής τα πράγματα δυσκολεύουν όταν μιλάμε για παράδειγμα για εκχώρηση μεγαλύτερων ε, μεριδίων ε, στους παραγωγούς των άλλων χωρών ή όταν λέμε ότι δεν θέλουμε εργασία, εργασία των παιδιών. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί αν θέσουμε αυτό, αυτή την πρώτη προδιαγραφή, αυτή την απέτηση θα πρέπει να γίνονται και έλεγχοι για να διαπιστώνουμε κατά πόσο τηρούνται. Αν γίνονται έλεγχοι θα πρέπει σε περίπτωση παραβίασης της ε, νομοθεσία να υπάρχουν και κυρώσει και από τι κυρώσεις ενδεχομένω να προκύψουν άλλα προβλήματα, όπου, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν εκ του νόμου προβλεπόμενες χειρώσει. Άρα πώς ε, θα προτείνουμε να τιμωρούνται κάποιες ε, τέτοιε διαδικασίε. Και να πω και κάτι άλλο. Εγώ έχω παιδιά και γόνια. Οι οποίοι α, α, αγοράζουν τα προϊόντα τους όχι ανάλογα με τις εντολικέ αρχές και τις ειδικές αρχές, αλλά αγοράζουν ό,τι είναι πιο φθηνό και ό,τι τους αρέσει πιο πολύ. Άρα, θέλω να πω ότι εσεί με την αγοραστική σα δύναμη μπορείτε να επηρεάσετε την κατάσταση. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Στη Γερμανία, ένα ε, πάροχος ε, τέτοιων προϊόντων κατηγορήθηκε για παιδική εργασία. Μπορούμε να πούμε ότι αρνούμαστε και απορρίπτουμε την κεντρική εργασία, αλλά πολύ απλά είναι ιστορικό φαινόμενο ότι σε κάποιε χώρε χρειάζεται η παιδική εργασία. Και υπήρχε και στη Γερμανία αυτό. Αν δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει η παιδική εργασία, α κάνουμε προτάσει για το πώ μπορεί να αποφευχθεί η παιδική εργασία. Και έτσι ο, ο, το έκανε μεγάλη προσπάθεια για να αποφύγει την παιδική εργασία, αλλά για να εξασφαλίσει παράλληλα ότι και τα παιδιά θα πήγαιναν στα σχολεία. Γιατί να μένουν μόνο του τα παιδιά δεν έχει νόημα, θα πρέπει κάτι να κάνουν να προκόψουν, να πάνε παραπέρα. Αυτά είναι λοιπόν στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο. Μπορούμε να κάνουμε προδιαγραφέ. θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, αλλά πιστεύω ότι αν εσεί, οι νέοι πείτε ότι κοιτάξτε, όχι, αυτό δεν το θέλουμε, αυτό θα είχε πολύ μεγαλύτερε συνέπειε από την επιβολή νομοθεσία και κυρώσεων. Σα ευχαριστώ και ω πρόεδρο τη Επιτροπή να πω και εγώ δύο λόγια. Όντω, στην Επιτροπή διαπιστώνουμε ότι μεγάλη είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων και θα πρέπει αυτό να συμπεριληφθεί στα δεδομένα και σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλε από περιοχές συγκρούσεων και σε ό,τι αφορά άλλους τομείς. Νομίζω ότι η καλύτερη η λύση είναι να είναι κοινή η ευθύνη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων, ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά να συνενωθούν σε ένα πακέτο και να κοιτάξουμε και τον έλεγχο τη εφαρμογής. Μιλήσαμε λίγο πριν για τη συμφωνία στον Παγκλαντές, όπου αυτό συνέβη ακριβώς. 220 εταιρείε που εισάγουν προϊόντα από τον Μπαγκλαντές με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν να είναι δεσμευτική και υποχρεωτική η επιθεώρηση των, εργασ... των εργοστασίων για να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι εργασιακοί όροι και να βελτιωθούν τα εργασιακά με ένα πιο σαφές σχέδιο ελέγχου. Αυτός είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι επιχειρήσεις με σαφή συστήματα ελέγχου. Ο λόγος και πάλι σε εσά. Η Έλεν, ίσως πρώτη. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα γερμανικά. Ήτανε θετικά αυτά τα οποία αναφέρατε. Τώρα μπορεί φυσικά να υπάρχει και μια ιδεολογική διαφορά μεταξύ ημών. Εγώ βλέπω ότι πολλές φορές είναι υπερβολική η πίεση στις επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να επικρατήσουν οι αξίες αυτές του ελεύθερου του δικαίου εμπορίου θα πρέπει εμείς να μεταλαμβαδεύσουμε καλύτερα αυτές τις αξίες, να υπάρξει και μια μορφή κατάρτισης προς την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι έγινε σαφές αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Άκουσα αυτά που ελέγχθηκαν ότι δεν είναι ε, εύκολο να τα περάσει κανείς αυτά με εθελοντική μορφή, αλλά αυτή τη στιγμή σε ένα από τα οχτώ σε ένα, από κάθε 8 καφενεία πολλούνται προϊόντα fair trade, το οποίο ήδη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ θα προτιμούσα φυσικά να πάω σε αυτό το καφενείο να πάρω τον καφέ μου. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό, όπως πάντα γίνεται, οι νέοι θέλουν να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση ώστε να υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση στα θέματα αυτά, ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι ένα προϊόν παράγεται κάτω από συνδίκες δικαίου εμπορίου ή όχι. Και επομένως να έχει την επιλογή από εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εστονικά φαντάζομαι. Θα μιλήσω αγγλικά όμως. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε. Και είναι εντυπωσιακό το να ακούσουμε τόσες πολλές απόψεις ανθρώπων που έχουν την ίδια άποψη με εμάς. Απλώς θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να σταθώ σε κάτι που είπε ο κύριος Βίνκλερ. Ήταν από τους λίγους ο οποίος βρέθηκε σε αντιπαράθεση κατά κάποιο τρόπο μαζί μας. Όλα αυτά είναι θέμα ερμηνείας. Εγώ εκτιμώ αυτό το οποίο είπατε για την ήπια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία μορφή όμως ήπιας δύναμης, όπως ε, έχουμε δει και στις διαπραγματεύσεις, το θέμα είναι τι, τι φρασιολογία χρησιμοποιούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όταν λέμε εμεί ότι πρέπει να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν κάτι, αυτό ήδη είναι μια μορφή παρουσίασης αυτών των θεμάτων σαν να είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο να υπάρξει μια ρύθμιση. Εμεί δεν πρέπει να μιλάμε για να υποχρεώσουμε τι επιχειρήσει να κάνουν κάτι. Θα πρέπει να τι ενθαρρύνουμε και να του δώσουμε τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν νομίζω ότι οι επιχείρησει χρειάζονται τόση πολλή παιδεία. Δεν είναι εναγνία σε σχέση με την επίπτωση των πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν νομίζω ότι αυτές οι εταιρείε θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο. Δεν θέλει κανεί. σω είναι η αφέλεια τη νεότητα αυτό που λέω. Νομίζω ότι πολλέ εταιρείε θέλουν να κάνουν να κάνουν κέρδη. Αλλά και το πώ θα κάνουν τα κέρδη είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό και για του εργαζόμενου εκεί. Δεν θέλουν μονάχα να πουλήσουν κάτι, θέλουν να κάνουν, να προκαλέσουν την θετική αλλαγή. Γι' αυτό θα ήταν πιο σημαντικό να ενθαρρύνουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα στι εταιρείε να είναι πιο βιώσιμε. Αυτό σημαίνει φυσικά και ένα κώδικα συμπεριφορά, αλλά συγχρόνω να υπάρξει και τέτοια ρύθμιση στην αγορά, ώστε οι επιχειρήσει που έχουν πιο βιώσιμε πρακτικέ να μπορούν να επιβιώσουν, να μπορούν να είναι κερδοφόρε και έτσι να υπάρξει ένα τρόπο κερδοφορία, ο οποίο είναι και τρόπο αλλαγή του κόσμου. Η παιδεία τώρα και η κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντικέ και απαραίτητε. Συμφωνώ με τον κύριο Σταρμπάτη ότι είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και για μας να καταλάβουν οι καταναλωτές ότι έχουμε την αγοραστική ικανότητα για να αλλάξουμε τις παγκόσμιες πρακτικές. Δεν ξέρω όμως τι μπορείτε να κάνετε εσείς ε, ως Επιτροπή Ίντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερο για να πλησιάσουμε τους ομόλογους μας, τους νέους και θα θέλαμε να έχουμε τη βοήθειά σας για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε τους ομολόγους μας, τους νέους δηλαδή, για το πόσο σημαντικό είναι να ζούμε βιώσιμο και να αγοράζουμε βιώσιμο. Ευχαριστώ, λέω Πράγματι, <clears throat> τα προϊόντα δικαίου εμπορίου Fair Trade ε, είναι παρόντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπαθούμε μάλιστα να προωθήσουμε την χρήση τους επίσης ε, να ε, είναι όντως προϊόντα τα οποία διασυνδέουν τον παραγωγό με τον καταναλωτή με διαφορετικό τρόπο. Το Fair Trade λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα και μας απασχολεί εδώ στην επιχείρησή μας ε, και το θέμα της ευθύνης των εταιριών και όλα αυτά. Υπάρχει στενή διασύνδεση ανάμεσα στη δικιά σας πρόταση και τη δουλειά που κάνουμε στο Κοινοβούλιο ε, και σας παρακαλώ να παραμείνετε στις θέσεις σας με την έννοια ότι θέλουμε να συνεχίσετε να μας πιέζετε, να πιέζετε τους βουλευτές. Το δεύτερο θέμα είναι εμπόριο για όλους, trade for all. Υπάρχει μια νέα εμπορική στρατηγική, την οποία δημοσίευσε το Σεπτέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μέσω της οποίας ε, προσπαθούμε να μετακινήσουμε λίγο τον ε, κέρσορα του εμπορίου και των εμπορικών συναλλαγών έτσι ώστε ε, το εμπόριο να γίνει πιο σύγχρονο, να είναι έτσι σύγχρονο για την ε, εποχή που ζούμε, κατάλληλο και επίσης να μετακινηθεί προς τις αξίες. Και αυτό μας απασχολεί πολύ εδώ στην Ίντα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην ε, ε Δεσποινίδα Williams. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει ένα πολύ καλό σύστημα, αποτελεσματικό, έτσι ώστε να καταγράφει τις γεωγραφικές ε, προελεύσεις. Ε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να προσθεθεί σε αυτό το επιτυχημένο σύστημα και η γεωγραφική προέλευση από χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής ε, και του Ειρηνικού. Θα πρέπει να βοηθήσετε τις ε, χώρες αυτές έτσι ώστε να αναπτύξουν ένα δικό του σύστημα ε, τέτοιων γεωγραφικών προελεύσεων και επισημάνσεων έτσι ώστε να διασφαλιστεί το εμπόριο για όλους. Οι γεωγραφικές ενδείξεις, όπως τα ξέρετε ίσως, ε, χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να ορίζονται κάποιες, ε, ε, κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα όπως είναι ας πούμε ε, το ζαμπόν της Πάρμας ή το παρμεζάνο ή διάφορα άλλα. Να ξέρουμε δηλαδή ακριβώς ότι είναι το αυθεντικό προϊόν. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο αναγραφόμενο στην ετικέτα προσελκύει τους αγοριστές. Θα πρέπει να προστατέψουμε μέσω αυτής της, ε, της ε, ε, επισήμανσης της γεωγραφικής, καινοτόμα προϊόντα, προϊόντα τα οποία προέρχονται από ειδικέ καλλιέργειες ή από φάρμες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι καινοτόμες και οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτές τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να συνεχίσουν ε, την δουλειά που κάνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προστασία λοιπόν. Επίσης, ε, ως η ανάπτυξη τη υπαίθρου και η σωστή γεωργική παραγωγή μέσω τέτοιων ε, κινήσεων. Μία πρώτη ύλη θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει ας πούμε τον καφέ της Γουινέας, ε, τον ειδικό μπλε καφέ της Τζαμάικα, ε, επίσης ε, το μαύρο ειδικό πιπέρι από το Τρινιδάδ και το μπάγκο. και αυτά είναι λίγα μόνο από τα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αυτήν την ε, γεωγραφική, αυτό το γεωγραφικό ε, στοιχείο. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί αυτή η πολύ σωστή αρχή του Trade for All. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα σας δώσω μια καλή δεύτερη ιδέα. Ε, συνήθως αναφερόμαστε σε άρση των ε, ε, εμποδίων των εμπορικών εμποδίων. Εγώ όμως θα έλεγα ότι θα πρέπει να αντιστραφεί η πορεία και θα ήθελα κάποιες, κάποια εμπόδια να υπάρξουν για ορισμένες περιπτώσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε κάποια βήματα έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην αποτελεσματικότητα, στη διαφάνεια και σε κάποιες άλλες αρχές οι οποίες ε, είναι πλέον απαραίτητες εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια στρατηγική η οποία ε, θα συμπεριλαμβάνει ισοδίκαια όλους. Κατά την άποψή μας ε, θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικοί εμπορικοί κανόνες ανάλογα με το εμπορικό επίπεδο της κάθε, της κάθε χώρας. Ε, ε, πιστεύουμε ότι οι κανόνες για όλους θα πρέπει να ε, γίνουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι θετικοί για όλους γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις στείνουμε με την πλάτη στον τοίχο κάποιους καλλιεργητές, παραγωγούς, κτηνοτρόφους ε, ή αλληλείς, γιατί ε, στις χώρες τους είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες παραγωγής. Θα πρέπει στις εμπορικές συμφωνίες να μην βάζουμε πάνω από όλα μόνο το δικό μας συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων. Αυτό σημαίνει trade for all, εμπόριο για όλους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στα όχι μόνο εμείς αλλά και οι εμπορικοί μας εταίροι. Ε, αυτό που ενδεχομένως, ενδεχομένως χρειάζονται οι εταίροι μας είναι μια μορφή προστασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρωτού ξαναδώσω το λόγο στους συναδέλφους. Θέλω να χαιρετήσω μια ομάδα από την ε, Κάτω Σαξονία, από την δική μου εκλογική περιφέρεια. Καλώς ήλθατε όλοι εδώ πέρα το θέμα της γεωγραφικής ένδειξης προέλευσης. Είναι ένα από τα θέματα που πραγματικά μπορεί να προστατεύσει τις τοπικές παραγωγές και αυτή η έννοια που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τύχη μίμησης και σε άλλες περιοχές του κόσμου, στην Αφρική, αυτό περιλαμβάνει και στη συμφωνία μας ακόμα και με το Βιετνάμ για τη γεωγραφική προέλευση όπου υπάρχουν και εκεί περιφερειακά προϊόντα τα οποία θέλουν και αυτοί να την προστατεύσουν. Επομένως αυτό είναι ένας τρόπος να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε τις περιφερειακού χαρακτήρα παραγωγές. Βίνκλα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την πρόταση για τι γεωγραφικέ ενδείξει. να την κάνουμε upload είναι δύσκολο βέβαια αυτό, γιατί είμαι από χώρη της Ανατολικής Ευρώπης. από τη Ρουμανία. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είμαστε 10 χρόνια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε μόνο μία γεωγραφική ένδειξη. Πολύ σημαντική. Να σας πω ότι αυτό που αναφέρατε προηγουμένω και αυτό που ανέφερα και εγώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ισχύ και η δύναμη τη εκπαίδευση ε, τη παιδεία θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για την ανάπτυξη του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων για να εξηγήσουμε ποια είναι τα πλανεκτήματα αυτού του συστήματος. Γιατί ξέρετε ότι δεν είναι όλοι υπέρ των γεωγραφικών ενδείξεων. Υπάρχει μια μεγάλη χώρα, η ΕΠΑ, που δεν συμφωνεί με τις ε, γραφικές ενδείξεις που λέει μπορεί να κάνει κανείς ε, σαμπάνια όχι μόνο στην καμπανία αλλά βάσει μια συνταγή. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Και πάλι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τρόπους συνεργασίας. Δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσει γιατί εσείς στη γενιά σας ξέρετε ότι ο κόσμος είναι δικτύωση και είναι δικτυωμένος. Η οικονομική λοιπόν συνεργασία αποτελεί έναν καλό αγωγό, ένα καλό όχημα για την ε, ανάπτυξη στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής κτλ. Και κάτι άλλο. Μπορούσατε να μιλήσετε τη γλώσσα σας, αλλά θα έπρεπε να το έχετε πει εκ των προτέρων, γιατί στο κοινοβουλίο μας έχουμε 24 επίσημες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η δική σας συμμετρική. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. για το δεύτερο αυτό στοιχείο που αναφέρεται, τη δεύτερη ιδέα. Όχι μόνο κατάργηση των εμπορικών φραγμών, αλλά και προώθηση τη περιφερειακής ανάπτυξης. Ναι, αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, γιατί φυσικά στις εμπορικές μας ε, σχέσεις κοιτάμε το πώς αναπτύσσονται τα πράγματα και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Κοιτώντας λοιπόν τις αφρικανικές ε, χώρες, είναι ασύμετρες οι συμφωνίες ε, ασφαλώς. Είναι επαρκώς ασύμετρε, μήπω κάποιοι τομεί θα πρέπει να προστατευτούν με καλύτερο τρόπο. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Αλλά είναι σαφέ ότι με χώρε διαφορετική οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούν να είναι ισότιμε ε, οι διαπραγματεύσει και οι συμφωνίε θα πρέπει να υποστηριχθεί η περιφερειακή ανάπτυξη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το εμπόριο μεταξύ των λιγότερων αναπτυσσόμενων χωρών. Χωρών του Νότου με χώρες του Νότου. Προκειμένου αυτή η, η ισορροπία, για παράδειγμα μόνο με την εμπορία πρώτων υλών από τις χώρες αυτές να καταρρευθεί. Να δοθούν πιο πολλές δυνατότητε απασχόλησης και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο κύριος Σόλτς, ναι, σας ευχαριστώ και εγώ να συνεχίσω από εκεί που το άφησες Μπέρντε. Αφαίρεση κάποιων εμπορικών εμπορίων, και δημιουργία κάποιων άλλων. Να δούμε λοιπόν ε, τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα παράγουμε στο μέλλον, πώς θα γίνεται η ανταλλαγή προϊόντων. Trade for all ε, και για το περιβάλλον. Το περιβάλλον το βάλαμε στην ε, συνθήκη του Παρισιού στο επίκεντρο. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς στέλνουμε τα εμπορεύματα ποια προϊόντα μπορούν να κινηθούν με την κυκλική οικονομία. Και σε θέματα γεωργικής παραγωγής, παραγωγής τροφίμων, ποια προϊόντα καλύτερα να κινούνται περιφερειακά μόνο. Να λεφθεί και αυτό υπόψη. Για θέματα προστασίας του καταναλωτή χρειαζόμαστε γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. ουσίες τέτοιες οι οποίες ε, χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Διάφορα στοιχεία τα οποία είναι άλληλα εξαρτώμενα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εκτάξουμε σε πολυμερέ επίπεδο, λιγότερε λοιπόν διμερεί ενδεχομένω συμφωνίε και πιο πολλέ πολυμερεί διαπραγματεύσει για κοινή διαμορφώση των κανόνων. Κύριος Μπούχνερ, ευχαριστώ και θα ήθελα Κυρία Ραμπ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί μιλήσατε για τα θέματα αυτά των διαφόρων μορφών εμπορίου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα αλλά και σε σχέση με, τη συμφωνία για για τα αγαθά του περιβάλλοντος που έχουμε κλείσει με την Κορέα εδώ. Περιλαμβάνονται και αγαθά τα οποία δεν απαιτούν μεγάλες επενδύσεις ώστε να παραχθούν. Όταν όμως παρέχει κανείς το ελεύθερο εμπόριο και ανοίξει την αγορά για επιχειρήσεις οι οποίες λόγω του μεγάλου αριθμού προϊόντων που έχουν και του μεγέθους μπορούν να έχουν καλύτερη παρουσία στην αγορά, τότε οι επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν πατήσει, δεν έχουν καμία ευκαιρία να επιβιώσουν. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για αυτή την περίπτωση, ποια είναι η σκέψη σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, λέγει ο Ο κύρος Σταρμπάτη. Να σας υπενθυμίσω ότι όλες οι αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες ξεκίνησαν με προστατευτισμό, με ισχυρή προστασία για τα προϊόντα τους. Και μου το λένε πάντα οι συνομιλητέ μου. Θα τους βοηθούσε πάρα πολύ να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Και θα τους βοηθούσε αν οι Ευρωπαίοι δεν πετούσαν, δεν κάναν dumping των πλεονασμάτων τους σε μας Κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τον ανταγωνισμό στις χώρες αυτές τις αναπτυσσόμενες. Αυτό είναι λοιπόν ένα σημείο το οποίο πρέπει να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας να κάνω την εξή παρατήρηση για τον προστατευτισμό έναντι του ελευθέρου εμπορίου. Αυτό που λέτε με κεντρίζει να πω το εξή, ότι υπάρχουν εμπειρίες με τη στρατηγική αντικατάσταση των εισαγωγών έναντι εξαγωγικής στρατηγικής. Έδειξαν οι μελέτες της πραγματικότητας ότι όλες οι στρατηγικές αντικατάστασης των εισαγωγών αποτυγχάνουν τελικά γιατί αυτό χρειάζεται να ορθώσει κανείς φραγμούς για να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία κτλ. Αλλά κάποιος ο οποίος έχει τέτοιους φραγμούς δεν μπορεί να περιμένει ότι αυτοί οι οποίοι θα αναπτυχθούν πίσω από τους φραγμούς θα είναι ανταγωνιστικοί, θα είναι αντιχωριστικές επιχειρήσεις. Οπότε κάποια στιγμή αυτή η εξέλιξη σταματάει. Και υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω μεταποίηση. Αν προστατεύονται τα προϊόντα αυτά, τότε χάνουν οι επιχειρήσει αυτές τη δυνατότητα διεθνούς, διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορούν να τα μεταπίσουν κάπου αλλού. Επομένως, προτού πούμε ότι είμαστε υπέρ ή κατά του να ορθώσουμε εμπορικούς φραγμούς για ορισμένα προϊόντα, θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ξέρω από, από τον Φρίντρικ Λίστα από το Πανεπιστήμιο της ε, Τιβίνγκης, ο οποίος θεώρησε ότι το η προστασία, η δασμολογική μπορεί να είναι ένα συνολικό προ... πρώτο εργαλείο για την ανάπτυξη. Αλλά ξέρω εγώ ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη χρονική διάρκεια. Φιέλνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πολιτική είναι σημαντικό στοιχείο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αντικρουόμενων συμφερόντων και την επίτευξη του αδυνατού. Uh, I think when we talk about trade policy, especially... Η εμπορική... πολιτική και η πολιτική που αφορά τις αναπτυσσόμενες είναι ένα πολύ προφανές παράδειγμα. Και διάφοροι συνάδελφοι. επεσήμαναν ότι οι χώρε αναπτυσσόμενε θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τη δική του παραγωγή για να υπάρχει σωστή ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι το εξή. Όταν εισαγαγονται οι δασμοί, αυτό γίνεται για να αυξηθεί η ιστορική τιμή των τροφίμων, προκειμένου να μπορέσουν οι γεωργοί να τα βγάζουν πέρα, για παράδειγμα, Α, με το επάγγελμά τους. Εγώ, ε, όταν το κάνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζω προβλήματα όταν αυξάνουμε τις τιμές των γεωργικών προϊόντων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνονται φυσικά και οι τιμές για τα τρόφιμα, το οποίο ασφαλώς αποτελεί πρόβλημα για τους φτωχούς. Κάποιοι διατείνονται ότι οι δασμοί για τα τρόφιμα είναι ουσιαστικά φόροι για τους φτωχούς. Εγώ και οι συναδελφοί μου προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο πιο χαμηλούς γίνεται τους, ε, τα τέλη, τους δασμούς για τα τρόφιμα. Και είναι δύσκολο όταν οι φτωχές χώρες αυξάνουν τις δασμούς στις δικές τους χώρες, στα δικά τους τρόφιμα, τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί αυτοί έχουν πιο πολλούς φτωχούς ενδεχομένω. Άρα, προσπαθώντας να βοηθήσει κανείς τους ε, αγρότες, μπορεί να πλήττει τους πιο φτωχούς σε σύγκρουση συμφερόντων. Πρόκληση, λοιπόν, κάτι που θα έπρεπε ασφαλώς να κάνουμε, είναι να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε δασμούς που θα έβλαπταν τις φτωχές χώρες. Είναι σωστή όμως και η ιδέα που προέβαλε ο Πρόεδρος για την περιφερειακή διαμορφώση όλων αυτών των εξαγών. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα σχόλια ενός λεπτού. Μάλλον να δώσουμε το λόγο για ένα λεπτό για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το feedback αυτό. Αναρωτιόμουν πόσα μέλη του Κοινοβουλίου είχαν υπόψη τους ε, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την, ε, ε, το άρθρο 145 της Συμφωνίας με τις Κάρι Φόρουμ, το άρθρο 16 της αντίστοιχης συμφωνίας. Για να λειτουργήσουν λοιπόν αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει διαρκώς να είμαστε σε επαφή μαζί του. και γι' αυτό λοιπόν έχει τόσο μεγάλε επιπτώσει σε θέματα γερικών ενδείξεων σήμερα. Κάτι άλλο. Κάτι που έγραψα στην εργασία μου στο Κολέγιο της Ευρώπης. Ήμουν στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια διπλωματία και ήθελα να αναπτύξω την ιδεολογία του Ρόντνεϊ για να δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό σήμερα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να μην επαναληφθεί η ιστορία. Ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν την επανάπτυξη τη Αφρική από πλευρά τη Ευρώπη. Θα πρέπει να κάνουμε τη διαφορά ω Ευρώπη. Ευχαριστώ, η Ελένα. Ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι που είναι τόσο έντονε οι αντιδράσει ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή για τις εμπορικούς φραγμούς, σε ό,τι αφορά την επενδυτική στρατηγική Investment for All. Είναι μεγάλη η πρόκληση προκειμένου όλα αυτά να μην διαμορφωθούν όπως επισημάνθηκε σε διμερές αγώνα επίπεδο, αλλά και σε πολυμερές επίπεδο. Η διαφορά δε μεταξύ ένα συστήματος βάση εισαγωγών και του ελεύθερου εμπορίου ή του ελεύθερου εμπάσχη περιπτώσει εμπορίου με κάποιες ε, ε που θα έδινε τις χώρες τη δυνατότητα να αναπτύξουν βιομηχανία και οικονομικό κλάδο είναι σαφής. Το trade for all, το εμπόριο για όλους, δεν θα πρέπει να ισχύει ως trade with the same rules, δηλαδή εμπόριο με ίσους όρους. Όχι. Εμπόριο των συμμετεχόντων φορέων. Όχι μόνο η παραγωγή, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορεί να γίνει trade for the poor, εμπορία για τους φτωχούς. Όλοι θα πρέπει να ωφελούνται. Γι' αυτό και ονομάζεται Trade for All και έτσι θα πρέπει να διαμορφωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κ. Βίνκλερ, ο πρόεδρος. Ε, όπως βλέπετε, οι, οι βουλευτές είναι αναγκασμένοι να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα αναλάβω τα καθήκοντα του πρόεδρου Μπεντ Λάνε και να ξεκινήσουμε τον τρίτο γύρο, στο τρίτο θέμα το δείτε σήμερα. Δεν χρειάζεται εισαγωγικά σχόλια και εξηγήσει. Καυτό θέμα ήταν και θα παραμείνει και θα δώσω το λόγο στον πλήρη. Καλώς ήρθατε και πάλι λοιπόν. Η δεύτερη μου ιδέα σήμερα πρέπει να ζητήσω περισσότερη συμμετοχή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει καταρχήν να δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο της TTIP. Οι ρυθμίσεις που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές και μετά όλες οι αλλαγές που θα γίνουν στις διαπραγματεύσεις. Επίσης θα ήθελα να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών για δημόσια διαβούλευση σε σχέση με την συμφωνία αυτή. Στο διάστημα αυτό θα μπορούν όλοι να δώσουν κάποιες ε, ιδέες βάσει των οποίων θα γίνει νέος γύρος διαπραγματεύσεων τότε μονάχα θα μπορέσει να προχωρήσει προς μια ναι ή ου ψηφοφορία αυτή η συμφωνία. Εγώ προσπάθησα να διαλευκάνω τι ακριβώς κάνει η TTIP, αλλά χρειάζεται να βασιστώ σε αποσπασματική πληροφορία και διαρροές. Το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς διαμείβεται, αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη καχυποψία για την TTIP. Οι πολυμερείς συμφωνίες όπως η TTIP έχουν μεγάλη σημασία για το τον Ευρωπαίο πολίτη και δεν πρέπει να κρύβονται από τα μάτια του ιδίω. Όταν εκατοντάδε Αμερικανικέ εταιρείε έχουν πρόσβαση στο κείμενο των διαπραγματεύσεων σε πραγματικό χρόνο. Με το να γίνουν πιο ανοιχτά αυτά τα πράγματα, θα διαβεβαιώσετε και την κοινωνία των πολιτών θα έχουν καιρό να εξετάσουν αυτήν την ε, συνθήκη προτού οριστικοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κείμενο περίπου 1600 σελίδων που έχει φτάσει στην κατάληξή του μέσα σε δύο μήνες. Αυτό δείχνει ότι δεν γίνεται διαπραγμάτευση προς όφελος των πολιτών, αλλά σε βάρος των πολιτών. Επειδή πιστεύω ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και ανα... ανησυχώ για την απογοήτευση που αυξάνεται μεταξύ των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ σας ζητώ να, γίνεται, δώστε έμφαση στην δημόσιο, δημόσιο χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, ακόμα και αν αυτό χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αν οι διαπραγματευτέ δεν χρησιμοποιούν χρόνο για να υπάρξει η εμπιστοσύνη από του Ευρωπαίου, μπορούμε να καταλήξουμε με έλλειψη συνθήκης. με καμία συνθήκη στο τέλο. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Βίγκλερ. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω τον περιορισμό χρόνου που έχουμε. Σα ζητώ και πάλι για δύο λεπτά μονάχα να μιλήσετε και τώρα η κυρία για να μα δώσει μια νέα πρόταση. Εγώ θα ήθελα να προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει στην Κομισιόν να υπάρξει ένα άρθρο που στη διαπραγματεύση που να δίνει την δυνατότητα στους νέους να εποπτεύουν τη συμφωνία αυτή με το να έχουν ένα μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή από όλε τι εμπορικέ συμφωνίε που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία με την Καραϊβική είναι η μόνη η οποία συνδέει του νέου με την εποπτεία και την παρακολούθησή του. Και επίση τι γυναίκε και τα παιδιά θα εξασφαλίσουν ότι τα ωφέλη αυτή τη συμφωνία προ αυτού θα ενισχυθούν. Αυτό μπορεί να γίνει και για την TTIP και για όλες τις μελλοντικέ συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το εμπόριο να είναι εμπόριο για όλους. Στο Φόρουμ και την Συμβουλευτική Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή όπου εκπροσωπώ το δίκτυο των νέων επαγγελματιών από τις χώρες ΑΚΕ, εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε δικαίωμα να θέλουμε να είμαστε πλήρη μέλη, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο δικαίωμα λόγου. Με τον τρόπο αυτό που θα πρέπει να δοθεί στου νέου, δυνατότητα να παρακολουθούν τι ενδεχόμενα αρνητικέ επιπτώσει των συμφωνιών εμπορικού χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά προσθέμενη αξία να έχουν μεγαλύτερη συνειδητοποίηση οι νέοι για τι εμπορικέ συμφωνίε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη για όλε τι περισσότερε θέσει απασχόληση και θα προστατεύσει του ανθρώπου και τον πλανήτη. Ω ερευνήτρια στον τομέα του εμπορίου, ξέρω ότι οι νέοι είτε είναι απόντε ή δεν αναφέρονται παρά μόνο αποσπασματικά στις εμπορικές συμφωνίες. Αλλά εμείς θα πρέπει να έχουμε σε στόχο να έχουμε μια πλήρη ε, ικανοποιητική και αμοιβαία και για τι δύο πλευρές συμφωνία την τύπα. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι δεν πρέπει να μείνουν εκτό μη Και έχοντα συμμετάσχει σε μια ακρόαση για τα θέματα αυτά, άκουσα πολλού νέου οι οποίοι είπαν ότι δεν θα δεχτούν την δυτή πώ έχει. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο στεναρή στο να εξασφαλίσει την ενεργή παρουσία των νέων μέσω τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την παρακολούθηση όλων των εμπορικών συμφωνίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε το εμπόριο είναι πράγματι για όλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Στρέφομαι στου συναδέλφου στη Μαρία Αρένα. Πολύ γρήγορα, σε σχέση με την πρόταση που μόλις υποβλήθηκε, νομίζω ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν είναι ακριβώς και περιοριστικά ε, εμπορικές συμφωνίες ε, ε, αφορούν ολόκληρη τη ζωή και όντως θα πρέπει να περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα στοιχεία και συμφωνώ με την άποψή σας για το θέμα αυτό. Νομίζω μάλιστα ότι το Κοινοβούλιο έχει πετύχει αρκετά πράγματα από την Κομισιόν όσον αφορά την διαφάνεια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο της πλήρους διαφάνειας ε, και ε, λέω ότι οι διασφαλίσεις πρέπει και εγγυήσεις να ζητηθούν από την Κομισιόν αλλά και από τα κράτη-μέλη γιατί αυτά ε, αναθέτουν εξουσίες στην και δικαιοδοτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς προσπαθούμε, κάνουμε τη δουλειά μας στο Κοινοβούλιο, αλλά ε, θεωρούμε ότι ε, μέσω της Κομισιόν θα πρέπει να ε, εμπλακεί και η κοινωνία των πολιτών περισσότερο. Δεύτερον, όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθέρων ανταλλαγών Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπος τέτοιων συμφωνιών ε, στους νέου, ε, στις γυναίκες, ε, στην απασχόληση, στην ισότητα των φύλων, βλέποντας ας πούμε γεωργικές συμφωνίες με την Αφρική, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των εργατών γη και δεν υπάρχει ανάλυση της επίπτωσης που έχουν αυτές οι συμφωνίες στις γυναίκες αυτές, ε, ε, ε, πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει κενό. Επίσης υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες οδηγούν σε μη βιώσιμες συμπεριφορές και αυτό θα πρέπει να το καταδείξουμε όχι γιατί δεν θέλουμε εμπορικές συναλλαγές αλλά γιατί θέλουμε βιώσιμες εμπορικές συναλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους μας για την παρουσίασή τους. Ολλανδικά, Ολλανδικά μιλάω. Γι' αυτό μάλλον χρειάζεται τα ακουστικά σας, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συμβολή σας και για τις ιδέες σας και με εντυπωσιάζεται ότι έχετε τέτοιες ε, καλές ιδέες και θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να σας παρατρύνω να συνεχίσετε να έχετε τέτοιες ιδέες γιατί και εμείς θα πρέπει να είμαστε σε επαφή με τους πολίτες, αλλά και εσείς θα πρέπει να είστε σε επαφή μαζί μας και να μας ενημερώνετε. Και εδώ έχω να σχολιάσω σε σχέση με τον πρώτο ομιλητή το εξή. Οι μεγάλες εμπορικέ αυτές συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές και είναι σημαντικό λοιπόν να συμμετέχει ο πολίτη σε τέτοιε μεγάλε εμπορικέ συμφωνίε. είπατε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες στις διαπραγματεύσεις. Ας κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Ας συζητήσουμε το πλαίσιο το οποίο θέλουμε να δώσουμε στους διαπραγματευτές προτού καν ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Προκειμένου να έχουμε μια εντολή από το λαό και όχι όπως στην περίπτωση του ΣΕΤΑ, μια συμφωνία η οποία διακρίνεται από μια έλλειψη διαφάνειας. Λάβαμε έκθεση από 455 εταιρείε στον Καναδά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλούν να καταψηφίσουμε την ΣΕΤΑ. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει αν είχαμε συζητήσει από πριν με τους πολίτες του τι επιθυμούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να σας ξαναδούμε. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριος Μπέχνερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω το θέμα της ε, διαφάνειας. Ε, πρόκειται για ένα από τα βασικά προβλήματα στις εμπορικές αυτές συμφωνίες. Δυστυχώς αυτό δεν αφορά μόνο το TTIP, αλλά θεωρώ και για την ε, TISA. Όπου πολύ βασικά στοιχεία παραμένουν άγνωστα. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αλλάξουμε εδώ στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι οι συμφωνίες αυτές αλλάζουν ε, την, ε, την πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας, την δημοκρατική μας καθημερινότητα. Νομίζω λοιπόν ότι ανακύπτουν ε, πολύ βασικά ερωτήματα και πιστεύω ότι η απογοήτευση που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί πολίτε πολίτες σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται ακριβώς με τα θέματα αυτά και να σας υπενθυμίσω και μια άλλη σκέψη η οποία ήδη εκφράστηκε στη Γερμανία πριν από κάποιο καιρό σε μια ημέρα 320.000 πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά την ε, ΣΤΙΤΙΠ και τη ΣΕΤΑ. Αυτό το αγνοούν οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται μια αγανάκτηση η οποία και κορυφώνεται χρειάζεται πιο πολύ διαφάνεια αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει μέλλον. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Σταμπάτη. Όντως η διαφάνεια είναι απαραίτητο θέμα. Ω τώρα όμω, να επισημάνουμε, καμία άλλη εμπορική συμφωνία δεν ήταν τόσο διαφανή από το TTIP. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτό έγινε αρκετά αργά μια όλη διαδικασία. Εγώ είμαι υπέρ της διάθεσης, ανοιχτής διάθεσης όλων των εγγράφων. Όλα θα πρέπει να είναι δημόσια. Για να ξέρει πραγματικά ο κόσμος τι είναι σημαντικό. Ιδάλλως προκύπτουν τέτοιες ιστορίες όπως το TTIP Leaks. Θα έπρεπε όλοι να ξέρουν τι περιλαμβάνουν αυτές οι συμφωνίες. Και για την κυρία Αρένα, για τη μελέτη επιπτώσεων. Αυτό φυσικά εξαρτάται από πολλά στοιχεία, αλλά το γεγονός ότι οι μεν ε, υπολογίζουν α, δυνατότητε ανάπτυξη και θέσει απασχόληση ό,τι αφορά το TTIP και κάποιοι άλλοι είναι κατά και θεωρούν ότι θα μειωθούν οι θέσει απασχόληση. Όλα αυτά είναι εικασίε. Και φυσικά, αν αλλάξουν αυτέ οι εικασίε, αλλάζουν και οι συνέπειε. Το μοναδικό που ξέρουμε σίγουρα, αγαπητοί συνάδελφε, είναι ότι το διεθνέ εμπόριο ανοίγει τα σύνορα και γίνεται πιο έντονο ο ανταγωνισμό. Και όταν είναι πιο έντονο ο ανταγωνισμό, υπάρχουν και απώλειε το καθοριστικό είναι ότι οι μεμονωμένες χώρες όταν ανοίγουν τα σύνορά τους θα πρέπει να έχουν και συνδευτικά μέτρα προκειμένου να μην συγκαταλεχθούν τελικά στους ε, χαμένους ε, της, ε, του διεθνούς ανταγωνισμού και μην έχουμε την εντύπωση ότι μόνο κερδισμένοι βγαίνουν. Όχι, βγαίνουν και χαμένοι. Η πολιτική για το κεφάλαιο, για την αγορά εργασία και όλα αυτά θα πρέπει να είναι ανοιχτά και να έχουν προσανατολιστεί στο άνοιγμα των αγορών. Ιδάλω μπορεί κανεί να σε καταλεχθεί στου ιτημένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλειμα του όλου του τελευταίου ομιλητέ. Ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα ποιο είναι ο ρόλο του εμπορίου στο γενικό πλαίσιο τη αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια αρνητική κατάσταση και εδώ τίθεται και το θέμα της διαφάνειας. Εγώ βρίσκω πολύ καλό που θέτετε αυτό το ερώτημα. Γιατί οι νέοι να έχουν απόλυτη αδιαφάνεια σε σχέση με την εντολή που δίνουν οι κυβερνήσεις τους για τις ε, διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΠ. Έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις παράλληλα ε, έχουμε δει διάφορε διαπραγματεύσει με τις ΗΠΑ. Η εντολή διαπραγματεύσεων είναι κάτι που είναι ηλικία 20 ετών και είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποιο απόρριτο χαρακτήρα. Είναι γνωστέ οι οικονομικέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ΗΠΑ, αλλά ακόμα και αυτή η εντολή δεν είναι δημόσια. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να υπάρξει δημόσια έκφραση άποψη. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους, ε, στις προσδοκίες αλλά και να καταπρίνουμε και τους φόβους των ανθρώπων. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια συμφωνία η οποία θα δώσει μια προσθέμενη αξία. Εδώ έχει σημασία να εστιάσουμε περισσότερο στην διαφάνεια και εγώ τονίζω ότι πρέπει να, να δημοσιευτούν τα στοιχεία για όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΠ. Ευχαριστώ, Λεόπρο ο Πιτ. Ε... Ευχαριστώ. Εξαιρετικό ήταν που άκουσα τις απόψεις σας γι' αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι ε, η TTIP ήταν ε, καλή συμφωνία ε, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία. Ε, το ζήτημα βεβαίως ήταν ε, η διαφάνεια και έκανε η Κομισιόν κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι αρκετό. Αυτό προσπαθώ να πω. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μία από τις πιο διάφανες υφιστάμενες συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες, αλλά παρόλα αυτά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Και, εν πάση περιπτώσει, το, εγώ αυτό που λέω είναι όταν να συμφωνηθεί ένα κείμενο να δημοσιεύεται, να δημοσιοποιείται και αυτό δεν γίνεται. Αυτό που λέμε είναι περίπου τι κάνει στους διάφορους γύρους διαπραγμάτευσης, ε, αλλά δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, δεν ξέρουμε ποια ήταν η πλευρά, ε, τι έλεγε η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Ε, δεν είναι απλώς γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Αμερική, αλλά νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια διαπραγμάτευση να δημιουργηθεί μια κοινωνική δημόσια εμπιστοσύνη. Πρέπει να είμαστε τίμη, έντιμη ε, μεταξύ μας και με τους ε, εμπορικούς εταίρους ε, και να τους πούμε ότι κοιτάξτε μόνο με διαφάνεια προχωράμε, τίποτα άλλο δεν λειτουργεί. Επίσης, αυτό που είπε η κυρία Ρενά, ότι θα πρέπει να δούμε όχι μονάχα το θέμα του εμπορίου, ναι, να δούμε και το θέμα των γυναικών και την ισότητα των φίλων και βεβαίως εγώ θα πω οπωσδήποτε να δούμε και το θέμα της υγείας, που είναι κάτι που με απασχολεί άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το feedback. Θα σας πω μια ιστορία σχετικά με το δίκτυο νέων επαγγελματιών της, από τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού. Πριν από δύο χρόνια ε, άρχισα να δουλεύω, στην, να συνεργάζομαι με τη DigiTrade ε, και είδα ότι λίγοι σαν εμένα δουλεύανε σε αυτές τις υπηρεσίες. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ήταν αναγκαίο να έρθουν σε επαφή με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις νέοι άνθρωποι από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού τρόπο αυτό μπορούμε να διευρύνουμε, να ενισχύσουμε την ενσωμάτωση και επίσης να δώσουμε και μια νέα πνοή ε, ε, και να μεταφέρουμε τα δικά μας προβλήματα. Ε, πιστεύω ότι είναι πολλοί οι Ευρωπαίοι αλλά και μη Ευρωπαίοι, δηλαδή προερχόμενοι από τρίτες χώρες που έρχονται και εδώ και θέλουν να σπουδάσουν και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για συζητήσεις. Σας ευχαριστώ θα σας διαβεβαιώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου είναι πάντα ανοιχτή σε νέες απόψεις, γιατί εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να είναι σε ανοιχτό διάλογο με τους Ευρωπαίους πολιτές και αυτό ακριβώς που ενδιαφέρει τους νέους θα πρέπει να το ακούσουμε και να το λάβουμε υπόψη και να το ενσωματώσουμε στις διαδικασίες διαπραγματεύσεων. Το θέμα αυτό της διαφάνειας όταν πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες δεν μπορεί να αποκλειστεί όπως γίνεται τώρα. Είναι σαφές ότι είναι απαραίτητη μια τέτοια διαφάνεια. Εμείς έχουμε αγωνιστεί ως Επιτροπή ε, Ίντα. Στο παρελθόν ήταν πολύ λίγες συμφωνίες στις οποίες είχαμε πρόσβαση οι λίγοι βουλευτές είχαν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά και τα έγγραφα αυτά για την TTIP. Θα ήταν σημαντικό να βρίσκονται και στο διαδίκτυο ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των λαών να γνωρίσουν περί την Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες σας για το Fair Trade, το εμπόριο για όλους, τις εμπορικές ε, Διαπραγματεύσει και συμφωνίε και ελπίζω θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Χρειαζόμαστε κριτική στάση από τους πολίτες της Ευρώπης για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κρατήσουμε το εγχείρημα της Ευρώπης, ένα εγχείρημα για τους λαούς και όχι να βρεθεί η Ευρώπη σε αδυναμία να ικανοποιήσει τι προσδοκίε των Ευρωπαίων. Πρέπει όλοι να εργαστούμε ώστε να μπορέσει να μείνει στο σωστό δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι λοιπόν περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία. οι διμερείς εμπορικές σχέσεις και ο έλεγχος της ε, Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Εδώ και καιρό το συζητάμε και με τους διάφορους εμπνεκόμενους φορείς. Αποφασίσαμε να καταρτήσουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Ο κύριος Μπορέλη είναι ο εισηγητής, ο οποίος και κατέθεσε έγγραφο εργασία, που θα αποτελέσει και τη βάση των συζητήσεών μας. Δεδομένη τη σημερινή κατάσταση, νομίζω ότι θα πρέπει να συλλογιστούμε πώς θα συνεχίσουμε με την Τουρκία. Και άκουσα σήμερα ότι η Τουρκία ανέστηλε τον διακοινοβουλευτικό ε, διάλογο μεταξύ τουρκικού και ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό αποτελεί άλλο ένα ορόσημο το οποίο μας καλεί να σκεφτούμε το πώς θα μπορέσουμε να κινηθούμε επικοδομητικά. Από εδώ και πέρα έχουμε μαζί μας μία σειρά εμπειρογνωμόνων. Έξι εμπειρογνώμονες Και μια και είστε και θα σα παρακαλούσα να τηρήσετε το χρονικό όριο των πέντε λεπτών χρόνο ομιλίας. Ιδάλλως δεν θα βγάλουμε πέρα. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Πέτη για πέντε λεπτά. Αγαπητέ Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη ε, δυνατότητα να συμμετάσχουμε σήμερα στην συζήτησή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η εμπορική σχέση με, το, ε, ε, με την Τουρκία. Ο Γενικό Γραμματέα θα έπρεπε να είναι εδώ, αλλά είχε δεσμευτεί να είναι παρόν σε μια άλλη εκδήλωση. 23 εκατομμύρια ε, γεωργοί εκπροσωπούνται από την ε, κόπα κοζέκα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να σας πω ότι μετά από 20 χρόνια ε, συνεργασίας με τις γεωργικές οργανώσεις και συνεταιρισμούς της Τουρκίας έχουμε μάθει πολλά όσον αφορά το εμπόριο με την ε, Τουρκία. Το 1998 υπήρξε μια ιδιαίτερη εμπορική ε, συμφωνία που αντιπροσωπεύει περίπου 2,5 δις ευρώ. Αυτή η συμφωνία ε, μας δίνει δυνατότητα συμμετρής πρόσβασης στην αγορά και Επίσης ε, ε, αναφέρεται σε δασμούς ε, της τάξης του και προϊόντα με ειδικού δασμούς που καλύπτουν περίπου το 40% των εμπορίων. Έχουμε ε, εξαγωγές οι οποίες στο 10% καλύπτουν γαλακτοκομικά προϊόντα και το υπόλοιπο είναι γεωργικά προϊόντα. Γι' αυτό ε, ενδεχόμενη πάυση συμφωνίας με την Τουρκία θα αποτελούσε πραγματικό σοκ για ορισμένους τομείς, κυρίως όσον αφορά το τομέα του βοήου κρέατος και τον γαλακτοκομικό τομέα. Ε, επίσης ε, πρέπει να σας πω ότι 200 με 300 ε, εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσε να είναι το κέρδος σε περίπτωση υλοποίηση πλήρους συμφωνίας με την Τουρκία και αυτό σύμφωνα με μια μελέτη τράπεζας. Πέρα από το θέμα των ε, δασμών, το θέμα της ένταξης Τουρκίας στην Τελωνιακή Ένωση θα πρέπει να έχει σαν στόχο και την ε, ε, βελτίωση του κεκτημένου, γιατί υπάρχουν και, οι μη τα μη δασμολογικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αρθούν, κυρίως όσον αφορά φυτοϊγειονομικά ε, προβλήματα, ε, κυρίως όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την καταγωγή των ειδών, όσον αφορά επίσης ε, την, αναπαραγωγική διαδικασία και τις εισαγωγές φυτών. Επομένως θα θέλαμε και τα κεφάλαια αυτά να ανοίξουν στις εμπορικές συζητήσεις με την Τουρκία. Μέχρι τώρα... 25%. Ε, ε, ε, της τιμής είναι, προέρχεται από στήριξη και το ίδιο συμβαίνει και σε ορισμένες άλλους τομείς όπως ας πούμε στον τομέα της ζάχαρης στην Τουρκία και είναι σαφές ότι εάν ανοίξουν οι τομείς αυτοί για την ζάχαρη ας πούμε θα αποτελέσει, θα αποτελέσει πρόκληση. Επίσης ε, κάνει κάποιες επιστροφές ε, η, η ε, Τουρκία και αυτό θα ισχύσει μέχρι το 2020 ε, και θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Ε, έχουμε την πρόσβαση στην αγορά ε, που οι προκλήσεις δεν είναι πολύ μεγάλες και επομένως για μας οι πιο μεγάλες προκλήσεις αφορούν τους μη δασμολογικούς τα, τα μέτρα τα οποία δεν σχετίζονται με δασμολογικά εμπόδια ε, αυτά θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και ευχαριστώ που δεν ξεπεράσατε το χρόνο σας. Η Ιζαμπέλ Βεϊλέρ από την Unitex. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα. Λέγομαι Ιζαμπέλ Βελέρ και ε, εργάζομαι στην Eurotex, η οποία εκπροσωπεί την Συνομοσπονδία κύκλος υφαντουργίας ε, και σχετικών μηχανημάτων. Να σας πω ότι εκπροσωπούμε 100 ε, τόσες ε, εταιρείες οι οποίες έχουν το 2015 69 εκατομμύρια τζίρο Κυρίως ε, οι μέλη μας ε, είναι οι, μη, ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς της κλωστοϊφαντουργίας. 44 δις ε, ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο αφορούν τη δραστηριότητά μας, ενώ 2,6 δις είναι η εξαγωγική δραστηριότητα ε, προς ε, την Τουρκία, 5,8% δηλαδή του μη ενωσιακού μας εμπορίου. Το ισοζύγιο είναι αρνητικό και τα τελευταία 10 χρόνια επιδεινώθηκε κατά 17%. Οι εισαγωγές Ε, ειδών ένδυσης ε, από την Τουρκία ε, αντιπροσωπεύουν 14 δις για το 2015 και καλύπτουν 44% της παραγωγής της, Ιταλίας, της Τουρκίας συγγνώμη, και αναφερόμαστε κυρίως σε σακάκια, παντελόνια, ρούχα ένδυσης για τις γυναίκες κυρίως. Μέχρι τώρα Έχουμε ε, επικεντρώσει την προσοχή μας σε τρία σημαντικά θέματα. Ε, το ένα είναι το καθεστώς εισαγωγών, το δεύτερο είναι ε, η τα μη τελωνιακά εμπόδια και το τρίτο είναι οι τιμές εισαγωγής. Όσον αφορά το πρώτο τμήμα και σχετικά με το ERF, αυτών των εντύπων λοιπόν καταχώρησης, θα πρέπει πριν από την εξαγωγή για πρώτη φορά να συμπληρωθεί ε, από την ε, χώρα ε, και ισχύει για ένα χρόνο. Επίσης, οι εξαγωγείς θα πρέπει να καταγραφούν στο e ΕΚΙΠ που είναι η τουρκική, ο τουρκικός οργανισμός για τις ε, εξαγωγές. Αλλά βεβαίως ε, κανείς δεν θέλει να αποκαλύψει ε, πολύ ευαίσθητες και απόρριτες πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποτελεί, εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις, είτε γιατί αντιμετωπίζουν αντιμετωπίζουν μεγάλο διοικητικό άκρο είτε γιατί ε, έχουν προβλήματα αποκάλυψης ε, ε, πληροφοριών. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που σας είπα για μη δασμολογικά εμπόδια. Εδώ υπάρχουν σημαντικά προβλήματα γραφειοκρατικά, όπου έχουμε διπλούς ελέγχους για λόγους ανείχνευσης χημικών ουσιών και ποιότητας. Δεν καταλαβαίνουμε πω αυτοί οι διπλοί έλεγχοι μπορούν ε, να ε, ελέγξουν την προέλευση των ε, υλικών και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν μεγάλες καθυστερήσεις στα τελωνία. Τέλος, ε, η αποστολή δειγμάτων ε, αποδεικνύεται πολλές φορές ε, πολύ, πολύ δύσκολη στην Τουρκία. Όσον αφορά τώρα τα, τις σχετικές, τα σχετικά μηχανήματα για την περίπτωση της Τουρκίας, η Τουρκία πρόσφατα αποφάσισε αύξηση των δασμών, αλλά το 2012 αναφέρθηκε ε, ο, ανέφερε μάλλον η Τουρκία ότι δεν θα ε, εφαρμόσει επιπλέον ε, δασμούς και βάρη για τα προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία και λόγω πολλών προβλημάτων συνεννόησης δημιουργούνται παρεξηγήσεις όσον αφορά τα δελτία προέλευσης ε, για προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας ε, προβλήματα και καθυστερήσεις. Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σας πω ότι η Eurotex εργάζεται σε εργαστή συνεργασία ε, με τις ε, τουρκικές ε, αρχές, είτε πρόκειται για τις οργανώσεις της βιομηχανίας, είτε τις μεταποίησης, είτε και των εμπόρων. Ζητούμε να αναλυφθεί δράση όσον αφορά πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία είναι δυσαπείλητα για την ώρα. Πολλοί συμφωνούν ότι οι ε, ε, προτιμήσεις οι οποίες αφορούν την Τουρκία ε, έχουν πλέον παλιώσει και επομένως θα πρέπει να ληφθούν κάποια νέα στοιχεία και κάποιες νέες αποφάσεις. Εμείς ε, δουλεύουμε σε συνεργασία στενή με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομάδα για τα κλωστοϊφαντουργικά ε, και στην ομάδα δράσης ε, για τις ειδικέ συμφωνίες για την κλωστοϊφαντουργία. Η Eurotex πρόσφατα ζήτησε από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, DigiTrade, να συμπεριληφθεί εκπρόσωπος από την Τουρκία ως παρατηρητής έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε λύσουμε τα ε, υφιστάμενα προβλήματα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σίσαρτ από την ΙΤΟΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Εργαζομένων θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να συμμετάσχουμε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την επιχειροποίηση της εμπορικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η ETUC, η Ένωση εργατικών ενώσεων εκπροσωπεί 89 συνομοσπονδίες εθνικές από 39 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Τουρκία έχουμε τέσσερα μέλη, την ε, ΔΙΣΚΙΣ, την Κέσκ την, ε, και άλλες. Αυτό, κάποιες από αυτές πρόσκειται στο ΑΚΕΠΕ και άλλες στο ΖΕΠ ή στο ΧΑΔΕΠ για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας η τωρινή συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα Τελωνιακής Ένωσης έχει ξεπεραστεί και πρέπει να βελτιωθεί. Και αν λάβουμε υπόψη τις τελευταίες, τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει τίποτα για την ε, διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος στην Συμφωνία Τελωνιακής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει αυτές τις αξίες γιατί αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στη συμφωνία με την Τουρκία και σε, όπως σε άλλες χώρες. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν στην Τουρκία πολλά θέματα τα οποία πρέπει να τηρήσουν όπως είναι και οι προδιαγραφέ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τα κοινωνικά θέματα. Υπήρχε μια ομάδα εργασίας για το κεφάλαιο 19 και για το κεφάλαιο 14, αλλά όλα αυτά δεν έχουν καρποφορήσει. Το να ένα κεφάλαιο για το βιώσιμο εμπόριο που αναφέρεται από τον εισηγητή στο εγγραφό του θα μπορούσε να βασιστεί με, με την συμφωνία με την Νότια Κορέα αλλά βελτιωμένη. Έχουμε τη ΣΥΤΑ και άλλες συμφωνίες που είναι σε συζήτηση. Αλλά η έμφαση να υπάρχει ένα δεσμευτικό εργαλείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου στην Τουρκία. Είμαστε σαφείς. Η ΕΤΟΚ και οι συνομοσπονδίες εμπορίου έχουν καταδικάσει απερίφραστα το, την απόπειρα πραξικοπήματος. Εγώ έχω πάει στην Τουρκία πολλές φορές από το 1963 ακόμα και στη συνέχεια ως ε, το 1993 μάλλον και έχω προσπαθήσει να καταλάβω λιγάκι την Τουρκία. Καταλαβαίνω το τραύμα το οποίο προεκλήθη από, αυτό το, από αυτήν την απόπειρα πραξικοπήματος. Η προσπάθεια αυτή η κατάλυση του συστήματος ιδίως από στρατιωτικές δυνάμεις για να Ανατσαπεί η δημοκρατία είναι ενέργειες που είναι πάντα απαράδεκτες. Ζητούμε όμως μια ανεξάρτητη ε, έρευνα και η απαραίτητο δίωξη αυτών οι οποίοι εμπλέκονται βάσει του γράμματος του νόμου. Αλλά επίσης εκφράζουμε και τις ανησυχίες μας για τις δραστικές ενέργειες της ε, τουρκικής κυβέρνησης αμέσως μετά την ήττα του πραξικοποιήματος. Αυτή τη στιγμή πάνω από 125.000 πολίτες κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και εργαζόμενοι, ακαδημαϊκοί ε, καθηγητές, ε, αστυνομικοί, τοπικές αρχές, ακόμα και επιχειρηματίες, ακόμα και εκλεγμένα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν βρεθεί στη φυλακή ή έχουν απολυθεί από τη θέση τους. 40.000 έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί. Υπάρχουν καταγγελίες για βασανιστήρια. Κατά την άποψη των μελών μας, είναι 46.000 άτομα που έχουν αναστα... έχει ανασταλεί η σχέση τους και έχουμε 76.000 άτομα τα οποία έχουν απολυθεί και αυτοί, αντίθετα με τους προηγούμενους που παίρνουν τα 2-3 του μισθού του, τους δεν παίρνουν απολύτως τίποτα, ούτε μία λίρα. Υπάρχουν πολυθεσμοί, μέσα ενημέρωσης, ενώσεις πολιτών, ιδιωτικές εταιρείες που έχουν κλείσει και έχουν κατασχεθεί τα στοιχεία ενεργητικών του. Αν δείτε την έκθεση τη Κομισιόν τη 9 η Νοεμβρίου, είναι ολε οι λεπτομερειε εκεί. Για λογου οι οποίοι μα φαίνονται απόλυτα αυθαίρετοι πολλε φορε που έχουν να κάνουν πράγματα που έγιναν πριν από 20 χρόνια. Η απόπειρα πραξικοπήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ω ένα πρόσχημα για να καταληθεί η δημοκρατία με ένα κράτο έκτατης ανάγκη στο διενετικές χωρί δημοσια χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο και έχουμε μεγάλη ανησυχία για το γεγονό ότι η κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει την θανατική ποινή. Τον Οκτώβριο η αντιπροσωπεία μας συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας αλλά και εκπροσώπους από ε, συνδικαλιστικές ε, ενώσεις που κατηγορήθηκαν ότι ήταν οπαδοί του Γιουλέν ή του ΠΚΚ. Χιλιάδες λοιπόν έχουν συλληφθεί από αυτούς. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε και είναι υπό εποπτεία. Προσπαθήσαμε λοιπόν μαζί με τη, τους, τα μέλη μας να παρακολουθήσουμε αυτή την κατάσταση. Δέκα μέρες αργότερα ήμουν στα Άδανα για ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν 200, 200 νέοι για το δείπνο ε, που έκλεινε την ε, διαδικασία αυτή. Του, του συνέλαβε, συνέλαβε λοιπόν η αστυνομία πάρα πολλά από τα άτομα αυτά χωρίς κανένα λόγο. Και αυτό για ενέργειε που θεωρεί ότι έγιναν πριν από δύο χρόνια. 24 Ιουλίου ετέθησε λειτουργία ο νόμο έκτακτη ανάγκη και έχει παραταθεί και φαίνεται ότι αντιβαίνει σε τρία νομικά εργαλεία τα οποία έχει υπογράψει η, η, η Τουρκία, η Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνε του Διεθνού Γραφείου ε, Εργασία κτλ. Η Τουρκία λοιπόν παραβιάζει το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί λοιπόν βιάζεστε εσείς για να επικαιροποιήσετε αυτή τη συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξετάσει και κλείνω, ναι, να παγώσουν οι διαπραγματεύσεις ένταξης και να εξεταστούν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης με την Τουρκία. Εμείς θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί, αλλά ελπίζουμε ότι θα λάβετε όλα, υπόψη όλα αυτά που λέμε. Ο κύριος Μπαχαντέρ, καλή αγασή από την τουρκική ε, Ένωση του ΣΥΑΤ των Τούρκων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών. Εμείς είμαστε μέλη της Business Europe, είμαστε τμήμα του συνασπισμού Β20 και εργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο. Γιατί, Γιατί οι περισσότερες εταιρείε μας Μάλλον συνεργαζόμαστε και με το εμπορικό επιμελητήριο τη Κίνα, γιατί πολλέ από τι εταιρείε μα που δραστηριοποιούνται στην Κίνα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θέλουμε να εξετάσουμε και αυτή τη διαδικασία εξυγχρονισμού. Η εκπροσωπεί περίπου 55 με 60% του ιδιωτικού τομέα στην Τουρκία και 80% των εξαγωγών μας καθώς και 85% των ε, φορολογικών εισόδων του τουρκικού κράτους. Έχουμε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ των μελών μας και υπάρχουν και εταιρείε ε, έχουν 100% τουρκική ιδιοκτησία και είναι δημόσιες εταιρείες ή επίσης εταιρείες οι οποίες είναι ξένης προέλευσης. Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ευρωπαϊκές επενδύσεις ή επίσης πρόκειται και για συμπράξεις με τουρκικές εταιρείες. Όλες εδώ αυτές οι εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία είναι μέλη μας και επομένως συμμετέχουν στις ενέργειές μας σε σχέση με τη διαμόρφωση απόψεων στην Τουρκία και μας έχουν υποστηρίξει από την αρχή. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Εδώ χρειάστηκε να αλλάξω λίγα την ομιλία μου. Το εμπόριο έχει συμβάλει πάρα πολύ στην, στο κοινό μας εγχείρημα στην αρχή, από την αρχή. Αλλά τώρα διατρεχούμε μια από τις πιο σημαντικές επιχει... Ε, χρονικές περίοδου όπου οι αξίες μας και οι συνεργασίες μας έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα μέσα στην κοινωνία μας για πολιτικούς λόγους αλλά και για τη νέα, με, μέσω της νέας βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιοποίησης. Στην Τουρκία βλέπουμε τα προβλήματα αυτά τα οποία εξετάζονται από εσά και πρέπει να αντιμετωπιστούν και πολιτικά σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν άρχισα να έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την προηγούμενη ιδιότητά μου ήταν τότε που γινόταν η συζήτηση για την Τελωνιακή Ένωση εδώ. Τότε υπήρχε θανατική ποινή στην Τουρκία, υπήρχαν πολλοί κοινοβουλευτικοί που ήταν στη φυλακή υποδίωξη, υπήρχαν προβλήματα ε, βασανιστήριων, απαγόρευση της χρήσης άλλων γλώσσων εκτός της τουρκικής δεν ήταν μια λαμπρή δημοκρατική περίοδος, αλλά από τότε και με την Τελωνιακή Ένωση μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 2000 υπήρξε πρόοδος και η Τουρκία έφτασε να ικανοποιεί σχεδόν απόλυτα τα πολιτικά κριτήρια της Κοπενχάγης. Αυτή τη στιγμή είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Ως εκπρόσωποι της PCR, εμείς είχαμε υποστήριξης αλλά συγχρόνω έχουμε αγωνιστεί για την δημοκρατία και το κράτο δικαίου στην Τουρκία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα να συνεχιστεί η διαδικασία εξυγχρονισμού τη Θελωνική Ένωση, όχι μόνο για την οικονομική ανόρθωση τη Τουρκία, αλλά για να έχουμε και καλύτερε συνθήκε για του εργαζομένου στην Τουρκία και να λάβουμε υπόψη και τις οικολογικές πρόοδους που γίνονται στην Τουρκία και στο μεταπληκτικό τομέα. και να προωθήσουμε το γενικό πλαίσιο του κράτους δικαίου, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να μιλάμε για επιχείρηση, δεν μπορούμε να μιλάμε για την πρόοδο της κοινωνίας μας και του πολιτισμού. Η Τουρκία, όπως ξέρετε όλοι, έχει μεταφέρει πάνω από το 50% του εκεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά και έχει γίνει μια διαδικασία <clears throat> αναδιοργάνωσης που οδήγησε στη φιλελευθερωποίηση των αγορών αγαθών που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. και έχει δεχτεί ορισμένα σημαντικά στοιχεία όπως είναι τα μέτρα κατά των κρατικών επιδοτήσεων και κατά του ντάμπινγκ. Ένα μεγάλο μέρος των εξαγών της Τουρκίας είναι μεταποιημένα αγαθά και θα ήταν καλό και για την τουρκική οικονομία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει και περαιτέρω φιλελευθερωποίηση. Είναι χρήσιμο να έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι σημαντικό να είμαστε πιο ανθεκτικοί, να έχουμε πιο υψηλά πρότυπα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και αυτό ισχύει επίσης και για τις δημόσιες προμήθειες που θα βελτιώσει το νομικό πλαίσιο στην ε, Τουρκία και θα οδηγήσει σε καθα... καθαρότερο τρόπο χρηματοδότησης πολιτικής και των δημοσίων αγορών. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν υψηλότερα πρότυπα με τα οποία πρέπει να συνάδουν αυτές οι διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, όπως ισχύει και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στην οικονομία της Τουρκίας. Έχουμε στα άλλα κεφάλαια, υπάρχουν θέματα για την εμπορική πολιτική, αυτό είναι το κεφάλαιο 4 για την Τουρκία και πρέπει ίσως να καταλήξουμε και σε, ένα νέο, σε μια νέα διάταξη που να συμπεριλαμβάνει περισσότερο την Τουρκία στην λήψη αποφάσεων. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο των υπηρεσιών 75% της οικονομίας της Τουρκίας βασίζεται σε αυτές και γι' αυτό είναι απαραίτητο ο τομέας των υπηρεσιών να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί χάρη σε αυτήν την, ε, τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακή ε, συμφωνίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει και πρόοδο στο νομικό πλαίσιο της Τουρκίας αν το ε, μοντέλο το οποίο θα ακολουθηθεί είναι αυτό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης που να έχει την απαραίτητη φιλελευθερωποίηση εάν αντίθετα ακολουθηθεί το σχέδιο του ΓΚΑΤ για τις υπηρεσίες, τότε δεν θα υπάρχει ένα πρόσφορο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο προτιμούμε. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα παράγοντα πρόοδου στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το να μην υπάρξει πρόοδο ή να παγώσουν οι σχέσεις μα, αυτό θα είναι κομμάτι του προβλήματος Θα είναι παράλογο να θεωρούμε ότι αυτό το οποίο ήταν κομμάτι του προβλήματο μπορεί να είναι κομμάτι τη λύση. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε μια λύση που θα είναι καλύτερη για όλου να προχωρήσουμε για την Τελωνιακή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Αιντίν. Σα ευχαριστώ πρώτα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη τη Επιτροπή ΣΥΝΤΑ που μα έδωσαν αυτή την ευκαιρία να πάρουμε το λόγο σήμερα. Οι τουρκικέ επιχειρήσει και η Συνομοσπονδία είναι βάση συμμετοχή σε θελούσια βάση εκπροσωπούμε 24 περιφερειακές ε, συνομοσπονδίες και διάφορες άλλες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Πάνω από 40.000 εταιρείε από όλη την Τουρκία. Η Κονφέντα αποτελεί το πιο ευρύ δίκτυο της των ε, τουρκικών δυναμικών επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων. Αποτελεί μια οργάνωση ευρωπαϊκών εταιριών με πάρα πολλούς απασχολούμενους. Και επίσης είμαστε σε στενή σχέση με την Business Europe και ως βασικός, βασική ε, εκπρόσωπος των τουρκικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρούμε ότι ο εξυγχρονισμός και η, η βελτιστοποίηση της Τελειωνιακής Ένωσης είναι κάτι απαραίτητο για να υπάρχει ε, μια καλύτερη σχέση μεταξύ των δύο μερών. Πιστεύουμε ότι για να πετύχουμε τον σκοπό αυτό η στρατηγική των διαπραγματευτών θα πρέπει να προσπαθεί να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα στο εμπόριο μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Τελωνιακή Ένωση και η Σχετική Συμφωνία του 1995 απέδειξε ήδη ότι η οικονομική ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και για τις τουρκικές και για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες καταρχάς μειώνοντας τα εμπόδια για την ε, είσοδο στο διεθνές εμπόριο και κατά δεύτερον δημιουργώντας ίσους όρους ε, μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεγαλύτερων ε, ομίλων. Σήμερα είναι νέες οι προκλήσεις στο διεθνές προσκήνιο και αυτό διαμορφώνεται από την ψηφιακή οικονομία, από τις μετατοπίσεις του διεθνούς εμπορίου. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να ενημερωθεί η Τελωνιακή Ένωση να προσαρμοστεί στις εξελίξεις και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα πρέπει να καταστεί πιο λειτουργική, πιο συνεκτική και πιο αποδοτική η Τελωνιακή Ένωση και για να δρέψουμε στο έπακρον τα πλέον εκτήματα και για τους Ευρωπαίους και για τους Τούρκους ε, πολίτες. Καλούμε τους ε, εκπροσώπους και των δύο πλευρών να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδιαιτέρως με ένα ειδικό κεφάλαιο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, να υπάρχει πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά εργαλεία από τις μικρομεσαίες. Να επιλύσουμε τις προκλήσεις που θα προκύψουν από την εξχρονισμένη Τελωνιακή Ένωση και να εφαρμόσουμε την αρχή Think Small, Act Small σε πρώτη φάση. Και τέλος, προκειμένου να είναι λειτουργική αυτή η συμφωνία, θα πρέπει να επιλύσουμε και το θέμα των θεωρήσεων που δημιουργήσει ένα βασικό εμπόδιο μη δασμολογικό, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι μια συμφωνία που θα λάβει υπόψη τα, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μας βοηθήσει να θέσουμε εκ νέου σε νέα βάση τι συνεργασίε μεταξύ ευρωπαϊκών και τουρκικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δούμε το θετικό αντίκτυπο της βαθύτερης οικονομικής ενσωμάτωσης που θα επηρεάσει και τις δύο πλευρές και την κοινωνία. Και αυτό θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα κοινό όραμα βάσει της ε, ευρύτερη διαδικασία ενσωμάτωσης τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και τέλο η κυρία Τέκιν από, τους, ε, από τι γυναίκε επιχειρηματίε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Άσλα Χάντακιν, ονομάζομαι και είμαι εκπρόσωπος της Κάκεντας των Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών της Τουρκίας. Κάγκεντέρ. Να σας πω δύο λόγια για την Τελωνιακή Ένωση και να σας πω και ποιοι είμαστε. Η Κάγκεντέρ, λοιπόν δημιουργήθηκε το 2002 από 37 αντικεκριμένες γυναίκες επιχειρηματίες στην Κωνσταντινούπολη και έκτοτε έχουμε παραπάνω από 300 μέλη. Ένα δις ευρώ και εκπροσωπούμε διάφορους τομείς της οικονομίας. τη φαντουργία, υγεία, επικοινωνίες, ψηφιακή οικονομία, τουρισμός, χημεία, δημόσιες σχέσεις και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν οι κλάδοι εκπροσωπούνται στο δικτύο μελών μας και το όραμά μας είναι να υπάρχει καλή εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική, στην, οικονομική πολιτική ζωή και στην κοινωνική ζωή. Προωθούμε λοιπόν την ε, επιχειρηματικότητα των γυναικών όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν αυτή την ε, γενικότερη οργάνωση που περιλαμβάνει την Ένωση Γυναικών ε, Επιχειρηματιών, τις γυναίκες επιχειρηματίες της Μεσογείου και άλλες ενώσεις. Και αυτό δημιουργεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για την καλύτερη πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών στην χρηματοδότηση, στην κατάρτιση, στα δάνεια. Και αυτό και με τις συνεργαζόμενες οργανώσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα λοιπόν θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας την Τελωνιακή Ένωση από την πτυχή της ισότητας των φίλων για να ακουστεί και η φωνή των γυναικών επιχειρηματιών. Στα πλαίσια της Τελωνιακής Ένωσης οι τομεί οι οποίοι δεν έχουν συζητηθεί και δεν έχουν συμπεριληφθεί είναι οι τομεί ουσιαστικά στους οποίους εκπροσωπούνται πιο πολύ οι γυναίκες, όχι μόνο στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια αριθμητικά στοιχεία, επιτρέψτε μου. Οι γυναίκες επιχειρηματίες, το ποσοστό ήταν 4,5 το 2004. Τώρα έχει φτάσει το 8% στην Τουρκία. Ξέρω ότι είναι ακόμα χαμηλό. 110.000 γυναίκες επιχειρηματίες αυτό συζητάμε. Αλλά κοιτώντα στην Ευρώπη, 29% το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών. 11,6 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Οι γυναίκε επιχειρηματίε, μεγάλο αριθμό, θα συμφωνήσετε όλοι. Και ω τώρα η Τελωνιακή Ένωση δεν περιλαμβάνει τι γυναίκε επιχειρηματίε και τι τομεί του οποίου εκπροσωπούνται ιδιαίτερω. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή σα. Και οι έρευνε καταδεικνύουν ότι 82% των γυναικών επιχειρηματιών στην Τουρκία είναι στον τομέα των υπηρεσιών. 40% εξ αυτών στις ε, εμπορικές πωλήσει. 70% έχουν μικροεπιχειρήσεις. Αυτό σας ε, δείχνει που θα πρέπει να εστιαστεί η συζήτησή μας ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες. Κοιτώντας την Ευρώπη, οι τομείς είναι η υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες, εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα των γυναικών επιχειρηματιών στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια άλλα αριθμητικά στοιχεία. 8,1 εκατομμύρια στην ε, Τουρκία είναι ε, μισθωτές. 41,8 είναι στην ε, γεωργία, 14,6 στην βιομηχανία και 43,7% είναι στον τομέα των επιχειρήσεων. Άρα, ό,τι συζητάμε εδώ στο Κοινοβούλιο σήμερα επηρεάζει τις γυναίκες που απασχολούνται στους τομείς αυτούς. Κοιτώντας την ευρωπαϊκή πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε και τα θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πόσο ε, επηρεάζουν την αναπτυξιακή ατζέντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία. Είναι σημαντικό να συζητηθούν οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Τουρκία και στην Ευρώπη λοιπόν σήμερα. Θέλουμε η συζήτηση λοιπόν αυτή να συμπεριληφθεί στη συζήτηση για την Τελωνιακή Ένωση όταν ενημερωθεί. Είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Μπορέλη Έχουμε καλούς εταίρους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπουμε σε μια ε, ενημερωμένη, ανανεωμένη τελωνιακή ένωση που θα έχει λάβει υπόψη και την άποψη των γυναικών επιχειρηματών και τον κλάδο της γεωργίας όπου δραστηριοποιούνται ιδιαίτερως οι γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας. Και τώρα ο, Μάξος και ο, εισηγητής μας και ο μάλλον ο κύριος Μπορέλ και μετά οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, από την παρουσίαση του, του εγγράφου εργασίας μας. Ε, ε, σήμερα ταυτοποίησαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το πάγωμα της, ε, της για την ώρα της διαδικασίας ε, ένταξης. Ε, αυτό βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τούτη την Επιτροπή η οποία συμμετέχει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Κοινοβούλιο. Το ε, έγγραφο εργασίας ε, νομίζω ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο γιατί κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε τα προβλήματα χωρίς όμως να χάνουμε το γενικότερο πλαίσιο. Και κατά αυτή την έννοια ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε όλου όσοι πήραν το λόγο σήμερα. Ε, σήμερα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να παρουσιάσει η Κομισιόν τον Δεκέμβριο στο Συμβούλιο την πρόταση εντολής για να δούμε αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ε, κατανοήσει και θα έχει αποδεχθεί τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ως εισηγητής ε, βεβαίως θα ενστερνιστώ την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που όπως σας είπα και προηγουμένως ε, προχώρησε, δήλωσε ε, ότι επιθυμεί την, ε, το πάγωμα της διαδικασίας ένταξης για την ώρα. Βεβαίως θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε σαφή θέση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ακριβώς να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σούστερ. Ναι, ναι, ναι. Excuse me. Κύριος συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έδινα το... θα σας άφηνα εσάς αν θέλετε. Ο κ. Παμπλεξ είναι ο μας τη, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ παρόντες. Αλλά... Αλλά επειδή και εγώ έχω την ίδια άποψη μαζί του, είναι πολύ εύκολο να παρουσιάσω τις απόψεις του, σαν να ήταν δικές μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκομένους εδώ που ήρθαν να κάνουν τις παρουσιάσεις τους. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι, που είναι απαραίτητο να το αναγνωρίσουμε, είναι ότι υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παγώσουν οι διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Αυτό όμω δεν σημαίνει πρέπει να σταματήσουμε τι εμπορικέ συζητήσει ή τι εταιρικέ σχέσει. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι εμπορικέ ε, συζητήσει για μια δυνατότητα να συνεχίσουμε την επαφή. Ακόμα είμαστε αλληλεξάρτητοι με την Τουρκία και πρέπει να συνεχίσουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε την αγορά με υποόρους επί τη βάση κάποιων αρχών και η Τουρκία μπορεί να βελτιώσει μπορεί να βοηθήσει να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία θέλει να εξυγχρονίσει την Τελωνιακή Ένωση, η οποία είναι πεπαλαιωμένη λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Το έχουμε δει σε πολλές φορές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Τελωνιακή Ένωση χωρίς το μηχανισμό αυτό επίλυσης διαφορών. Αυτό είναι κεφαλαιόδες και πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό να διευρύνουμε αυτή την συμφωνία σε τομείς όπως είναι η γεωργία, οι δημόσιες προμήθειες, οι υπηρεσίες, βιώσιμη ανάπτυξη, μικρομεσαίε επιχειρήσει και φυσικά και η προστασία του περιβάλλοντο, βλέποντα τι γίνεται πρόσφατα στην Τουρκία. Είναι σημαντικό επίση να αναγνωρίσουμε ότι δεν πρέπει να δούμε μονάχα αυτά τα οποία ωφελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ασυμμετρία σε αυτέ τι διαπραγματεύσει που είναι πραγματικά ένα στοιχείο αδικίας και το λέω παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι Ευρωπαίος. Εμείς μπορούμε να αποφελθούμε από την Τελωνική Ένωση, αλλά η Τουρκία δεν μπορούν να υποφελθούν από αυτά τα στοιχεία της συμφωνίας. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι κάτι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος μου και γι' αυτό θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι, ότι φυσικά έχουν, ε, έχουν υποχωρήσει ορισμένα πάντα, έχουν μειωθεί σε σχέση με την ε, αρχική πρόθεση και γι' αυτό πρέπει να κάτσουμε και να βρούμε πάλι λύσεις επί τη βάση του κοινού συμφέροντός μας και γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνει η αναβάθμιση αυτής της θελωνιακής συμφωνίας. Ο κύριος Σούστερ. Και ο δικός μας κύριος δεν είναι εδώ. Και γι' αυτό θα μεταφέρω τη δική του ε, άποψη, αλλά στα αγγλικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τη χρήσιμη συνεισφορά τους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά έτσι ώστε να έχουμε καλές εμπορικές σχέσεις με την Άγκυρα στα πλαίσια ενός ανανεωμένου εργαλείου. Με μεγάλη πλειοψηφία ε, υπερψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα το πάγωμα, μέσω ψηφίσματος λοιπόν, το πάγωμα της διαδικασίας ένταξης. Ε, αυτό είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλουμε ε, να στείλουμε σε μια χώρα η οποία ε, έχει από, ε, από πολύ καιρό ήδη εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχει σε αυτή την κοινότητα, η οποία όμως μη είναι και κοινότητα αξιών. Ε, είναι εποφελής και προς τις δύο πλευρές οι οικονομικές σχέσεις και εμπορικές επαφές μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να εκσυγχρονίσουμε το εργαλείο της Τελωνιακής Ένωσης ε, το Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους ιδίως της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, να ενεργήσουν έτσι ώστε να διασφαλίσουν την, τον σεβασμό των οικονομικών και κοινωνικών προτύπων στην Τουρκία. Έχω και μία ερώτηση. Σύμφωνα με μία μελέτη ε, την οποία ε, ε, πρόσφατα δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Τουρκία συμμετέχει κατά 3,1% στις εισαγωγές γεωδιατροφικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ακόμα περισσότερο όσον αφορά το ποσοστό ε, είναι ακόμα πιο σημαντικό, δηλαδή 2,9 από αυτά τα 3,1 αντιπροσωπεύονται από το, ε, από το βόλιο κρέας και από το, τα, το κρέας προβάτων. Ε, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γεωργικό τομέα στι επαφέ μα και δεν πρέπει να το λησμονήσουμε. Αυτό ευχαριστώ κύριε Φτώχη. Τρει παρατηρήσει ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλο. Ε, συμφωνώ με του συζητητέ, τον κύριο Φιέλνερ και τον κύριο Σούστερ. Η συμφωνία θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Και για τι δύο πλευρέ είναι παροχημένη πλέον. Στά και αυτό. Και αυτό θεωρώ ότι θα ήταν και ευνοϊκό και γόνιμο αν γινόταν. Δεν αμφισβητείτε, Δεύτερη παρατηρήση για την Τουρκία. Η Τουρκία χρειάζεται πιο στενέ σχέσεις, θεωρώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη αγορά. Η μεγαλύτερη φαντάζομαι για την Τουρκία. Και η Τουρκία πρέπει να κάνει τη μετάβαση από εξαγωγέα πρώτων υλών σε, χώρα που μετά για τις πρώτες ε, ύλες. Και αυτό το όριο δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει η Τουρκία χωρίς ε, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι μεγάλος μοχλός. Ε. Τρίτο στοιχείο, πολιτικό περιβάλλον, πολιτική ατμόσφαιρα. Αυτά που θεωρούμε όλοι οικονομικά επωφελή, οικονομικά είναι πολιτικός πώς αμφισβητούμενο. Πολιτικός ε, απομακρύνεται η Τουρκία από τις αξίες τις οποίες θεωρούμε σημαντικές. Αυτό που είπατε μόλις ε, για την διακοπή των ε, διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας είναι σε μια πορεία σύγκρουση στην Τουρκία. Αν ρωτιόμαστε λοιπόν αν συνεχίσουμε να δεν πραγματευόμαστε business as usual, μήπως θεωρηθεί αυτό ως τάση ε, υπαναχώρησης. Στάση υπαναχώρησης είναι κριτική αυτή που έχει ασκηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το λέω αυτό με πάσα συνείδηση στους εκπροσώπους της τουρκικής οικονομίας οι οποίοι ήταν πολύ διαφωτιστικοί στις παρουσιάσεις τους. Θα πρέπει να φροντίσετε στις χώρες σας όμως να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το οικονομικό σε εύλογο. Γιατί αν συνεχίσουν τα πράγματα όπως ως σήμερα, το οικονομικό εύλογο δεν θα επικρατήσει υπέρ της πολιτικής πραγματικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σχάκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εκτιμώ την ευκαιρία να πάρω το λόγο για την ανάγκη ενημέρωση τη της Ένωση με την Τουρκία και πάλι. Ήταν πολύ επωφελή συνταλλαγή απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι καλό που ακούμε για του εμπλεκόμενου φορεί. Αλλά θεωρώ ότι ήταν αρκετά α, γρήγορα τα πράγματα και χρειάστηκε να βιαστούν. Αυτό να το έχουμε υπόψη και για την επόμενη φορά, γιατί θέλουμε πιο πολλά να μάθουμε από αυτού. ορίζω το γεγονό ότι προγραμματίζεται αποστολή το Δεκέμβριο στην Τουρκία για να μιλήσουμε με του διάφορου ε, Εμπλεκόμενε φορές Το είπαν και οι πιο πολλοί όσοι πήραν το λόγο τώρα. Το εμπόριο βάση κανόνων και η ενημέρωση των κανόνων είναι σύγχρονοι κανόνες, είναι κάτι απαραίτητο. Και όπως είπε ο εισηγητής, τους καιρούς που διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην λαμβάνουμε υπόψη και το ολοπολιτικό συγκείμενο στο οποίο συζητιέται η ενημέρωση της Τελωνιακή Ένωσης. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ψήφισε να παγώσουν οι σχέσεις με την Τουρκία λόγω παραβιάσεις ε, του κράτους, ε, παραβιάσεων του κράτους δικαίου. Οι απαντήσεις δε ότι πρόκειται για μια λαϊκίστικη φωνή και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μη νόμιμο θεσμικό όργανο δεν βοηθούν. Όταν πρόκειται σε, για εμπορικά ζητήματα, να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε, έχουμε πλήρη συνομοθετικά, συνομοθετικές αρμοδιωτές. Μα, ανησυχεί η κατάσταση στην Τουρκία, αλλά πιστεύω ότι πάντα καλό είναι να είμαστε σε άμεση επαφή και νομίζω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να συνεχίσει το έργο της και να Έχουμε υπόψη ότι η ενημέρωση ενός τόσο πολύπλοκου νομικού κειμένου όπως η Τελωνιακή Ένωση δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αρπακόλα. Θα πρέπει να δούμε και τι πολιτική βούληση υπάρχει για την διεξαγωγή της άσκησης αυτής. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή το Δεκέμβριο στην Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ, ο Helmut. Θα είμαι σύντομο, γιατί ακούσαμε και πολλά από τους συναδέλφους. Και βεβαίω ε, όλοι είπαν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πολιτικό πλαίσιο και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε ε, και για επικαιροποίηση, για εξυγχρονισμό, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, αν μιλάμε από πολιτικές ε, για την έννοια του trade for all, ε, εμπόριο για όλους, τότε θα πρέπει το εμπόριο να κάνει καλό, να είναι εποφελές και προς τους πολίτες και θα πρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη διάσταση του εξυγχρονισμού σε αυτό το θέμα. Η απόφαση της Ολομελίας της προηγούμενης εβδομάδος είναι σαφής και δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν υπάρχει τώρα αυτή η, αυτή δύναμη που μπορεί να οδηγήσει προς την ε, ε, αλλαγή. Και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη και επομένως πώς θα πρέπει να συνεννοηθούμε, να μιλήσουμε με τους εταίρους μας και βεβαίως ε, χαίρομαι που είχαμε εδώ σήμερα εκπροσώπους ε, της οικονομίας, της βιομηχανίας, είχαμε εκπροσώπους ε, των γυναικών, γιατί μέσω αυτών θα περάσει το μήνυμα ότι το πολιτικό πλαίσιο δεν είναι ακόμα κατάλληλο έτσι ώστε να υπάρξει ενημέρωση επικαιροποίηση της κατάστασης. Σύμφωνα απόλυτα με τον προλαλήσαντα αυτά που είπε ο κύριο Σόλτ και ο κύριο Σταρμπάτη. Η δική μου ερμηνεία τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα το ερμηνεύω κάπως διαφορετικά γιατί ελέγχθη ότι το εμπόριο είναι σημαντικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Θα πρέπει να δούμε στο γενικό πλαίσιο που βρίσκονται οι δυσκολίες στη σχέση μας με την Τουρκία. Γνωρίζετε εξάλλου ότι ο, ο τουρκικός στρατός έχει βομβαρδίσει χώρους οι οποίοι προστατεύονται από την UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά. Χώρους που είχαν ανθρώπους μέσα, οι οποίοι σκοτώθηκαν, πολλοί από αυτούς. Υπάρχουν φυλακές όπου βασανίζονται ιδίως οι γυναίκες. Έχουμε λοιπόν πολλά στοιχεία στην Τουρκία που δεν θέλουμε πιστεύω να τα ανα, ανταμείψουμε με μία ε, αναβάθμιση των εμπορικών μας ε, σχέσεων. Νομίζω ότι αντίθετα πρέπει να δώσουμε το αντίθετο μήνυμα. Φερό. Κοιτάξτε, εγώ ακούω μία συζήτηση η οποία είναι σουρεαλιστική. Γιατί ε, την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε το πάγωμα της διαδικασίας με την Τουρκία. Διαπιστώνω ότι σήμερα η Τελωνιακή Ένωση ε, ε, αναφέρει σαν προϋπόθεση ας πούμε την ένταξη της Τουρκίας. Θεωρώ ότι τούτη εδώ είναι μια πολύ καλοπροαίρετη έκθεση που αναφέρεται μόνο στα συμφέροντα της Τουρκίας. Η θέση μου είναι απλή. Εγώ θα ήθελα, όπως κάναμε στην περίπτωση του παγώματος της της διαδικασίας ένταξης θα ήθελα να σταματήσει και η διαδικασία για την Τελωνιακή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία, τα λέω αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν στέκει καλά ε, και γιατί πιστεύω ότι η Τελωνιακή Ένωση ε, Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα είναι μία επιπλέον απειλή. Και αυτή τη στιγμή η Τελωνιακή Ένωση με την ε, Τουρκία απειλεί άμεσα την γεωργία μας και θεωρώ ότι σήμερα σε μια χώρα η οποία έχει κόστος παραγωγής 50% τουλάχιστον χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος παραγωγής της Τουρκίας θα ήταν αυτοχειρία να με αυτήν την συμφωνία. Ο κ. Μαυρίδης. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο σημεία θα ήθελα να θίξω. Ε, ένα που θα αφορά τον εισηγητή. Πολλές εκθέσεις έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες ε, σε σχέση με την... And they go through a lot of suffering. I like to get a comment on that. Uh, ε, σχετικά με, άσκηση βίας ε, και ε, καταχρήσεις εναντίον παιδιών, κυρίως δε προσφυγόπουλων. καταλαβαίνετε εδώ λέω και την προσωπική μου άποψη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι δυνατόν να μην μας επηρεάσουν για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να στείλουμε πολιτικό μήνυμα στην Τουρκία, ε, κυρίως για να παγώσουν κεφάλαια και όχι έτσι ώστε να σταματήσουν αρχίσουν επισήμως ε, όλες οι διαπραγματεύσεις. Το είπα λοιπόν αυτό. Αλλά στο βαθμό που ίσως εκφράζω την πλειοψηφία των συναδέλφων, μπορώ να πω ότι αυτοί που ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα το πάγωμα κάποιων κεφαλαίων, μεταξύ αυτών και εγώ, ε, ξέραμε πολύ καλά ότι το πάγωμα αυτό ήταν γιατί ε, η το καθεστώς Ερδογάν ε, έχει αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και επομένως δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουμε συμφωνία που θα άγγιζε και θα επιλέγει και το, εμπόριο. Η Επιτροπή για Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα περιοριστώ στα όσα έχουν να κάνουν με την Τελωνιακή Ένωση και την εξυγχρονισμό αυτής. Όπως ξέρετε, μετά την ε, εκκίνηση των ε, προετοιμασιών το Μάιο του 2015 για την εξυγχρονισμό της Ελληνικής Ένωσης και από τουρκικής και από ευρωπαϊκής πλευράς, γίνονται προετοιμασίες για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό. Από πλευράς μας, φυσικά, όπως σε κάθε εμπορική διαπραγμάτευση, αυτό περιλάμβανε και την διεξαγωγή μελέτη αντικτύπου. Η μελέτη αντικτύπου αυτή υποδεικνύει με σαφήνεια ότι η Τελωνιακή Ένωση και η ενημέρωση αυτή θα ήταν αμοιβαίω επωφελή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Τουρκία. Θα εξυγχρονίζε το διμερές πλαίσιο διεξαγωγής εμπορίου και νομίζω ότι ακούσαμε πολλά παραδείγματα για διάφορες αδυναμίε σήμερα το απόγευμα της τρέχουσας Ελληνικής Ένωσης και η μελέτη δικτύπου που καταδεικνύει ότι τα ωφέλη θα περιλαμβάνουν όλους τους τομείς που ερευνήθηκαν στο τομέα το γεωργικό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ασύμμετρες σχέσεις στην παρούσα φάση εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ε, φιλελευθεροποίηση. Επίσης, ε, καλύφθηκαν διάφορα ζητήματα τα οποία τονίστηκαν και υπογραμμίστηκαν σήμερα το απόγευμα και τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε ό,τι αφορά την μέλουσα έκδοση της Τελωνιακής ε, ε Συμφωνίας. Αναφέρθηκε και βιώσιμη ανάπτυξη αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να προσταθούν στις διμερείς μας συμφωνίες, διατάξεις για τα κοινωνικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Προδιαγραφές και διατάξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό ακούστηκε και είναι πάρα πολύ σημαντική πτυχή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τελωνιακή Ένωση και τον εξυγχρονισμό της Συμφωνίας όπως ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση του 2016 για την πολιτική για την διεύρυνση, τη λάβατε πριν από κάποιες εβδομάδες, είναι στη φάση της οριστικής διαμορφώσης στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο από τους εμπεριογνώμονες για να απαντήσει. Ένα λεπτό σας δίνω το λόγο, εάν τον επιθυμείτε ασφαλώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιας και τέθηκε ερώτημα για ισορρευτικό αντίκτυπο στο εμπόριο και στην γεωργία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ψάξαμε και επιδιώξαμε μια προσέγγιση ελευθέρου εμπορίου. Αλλά αυτό που θα θέλαμε να εκτιμήσουμε σε ό,τι αφορά το εμπόριο με την Τουρκία είναι ε, θέματα μεσογειακών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, για παράδειγμα και θέματα εμποδίων που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τα φυτοπροστατευτικά. Αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και γι' αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο εμπορικός αντικτύπος της συμφωνίας στην γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Θα ευχαριστήσω λοιπόν τους εμπειρογνώμονες μας σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και η επόμενη ανταλλαγή απόψεων βάσει του σχεδίου της έκθεσης θα λάβει χώρα στις 26 Ιανουαρίου. Και αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της δημόσιας ακρόασής μας. Θα κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα για να βγουν όσοι δεν είναι συντονιστές.